Okay. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη και έχουμε και τους συντενιστές που θα συνεδριάσουν στις 6. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε γιατί μέχρι τις 6 πρέπει να έχουμε τελειώσει. Θα εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. με κάποιες αλλαγές. Γιατί ο κύριος Κάσπαρη στο σημείο 7 στην εμπορική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 25 του κύριου Γκότλιφ για το Διεθνές Εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ζητήσει και οι δύο μια μικρή αναβολή. Τα θέματα λοιπόν αυτά δεν θα συζητηθούν σήμερα. Έχουμε και το αίτημα του κυρίου Dartmouth για το 15. Η χορήγηση εγγύησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα τα πούμε αυτά σε νέα Ευρωπαϊκή. Finally, following a request by Mrs. who will not be available. Και η κυρία Σαρνές, Δεσαρνές δεν είναι ε, διαθέσιμη σήμερα. Άρα λοιπόν τα 22 και 23 θα αλλάξουν σειρά. Το 23 θα συζητηθεί τελευταίο αύριο το πρωί και το 22 θα είναι το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε αύριο το απόγευμα. Με αυτές λοιπόν τις μικρές αλλαγές στην ημερήσια διάταξη την εγκρίνουμε αρκεί να μην υπάρχουν από μέρους σας. Να πω και δύο λόγια για αυτές τις αναβολές, οι οποίες είναι αρκετά πολύ άριθμες και δεν ε, επηρεάζουν μόνο την ε, συνάντηση τη σημερινή, αλλά και τις επόμενες συνεδριάσεις μας, οι οποίες ήδη έχουν και αυτές πολύ φορτωμένη μερίσια διάταξη. Λαπώ λοιπόν πως θα πρέπει οι αναβολές αυτές να αποτελούν την εξαίρεση, γιατί από τη στιγμή που έχει εγκριθεί το σχέδιο μερίσιας διάταξης, θα πρέπει οι εισαγητές να εξασφαλίζουν πως θα είναι διαθέσιμοι όταν θα συζητάμε τις γνωμοδοτήσεις τους. Ελπίζω λοιπόν μετά από αυτά οι συγητές και οι συντονιστές και οι υπόλοιποι από εσά να με ακούσουν και να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου είδους περιστατικά. Περνάμε λοιπόν στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 28 και 29 Σεπτεμβρίου, το σημείο 2. Εγκρίνονται λοιπόν εφόσον δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις ή σχόλια μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Σήμερα και αύριο στις συνεδριάσεις που θα κάνουμε ε, θα έχουμε και τη δυνατότητα να ακουστούμε μέσω web stream, εκτός βέβαια από το κομμάτι που είναι και κλεισμένο των θυρών. Σας έχει μοιραστεί και όλο το σχετικό υλικό. Αύριο για το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας, να σας πω πως θα συνεδριάσουμε σε μια άλλη αίθουσα, όχι εδώ, Στο ESP 5G2 χρειάστηκε να επαναπρογραμματιστούν αρκετές συνεδριάσεις λόγω των πλημμυρών που είχαμε στο άλλο κτίριο. Έλαβα και μία επιστολή. Sullivan Έλαβα λοιπόν την επιστολή αυτή από τον προηγούμενο διευθυντή, την προηγούμενη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης για το εμπόριο που μου έστειλε κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις και πρέπει να πω ότι έχει διοριστεί από τη Βαρόνη Άστον ως ε, Γενική Διευθύντρια της Νέας Υπηρεσίας για τις Εξωτερικές Σχέσεις. Φεύγει λοιπόν από την DigiTrade και μου ζητά να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής μας για τον επαγγελματισμό και τη στήριξη με την οποία εργαστήκατε σε θέματα εμπορικής ε, πολιτικής από την αρχή της θητείας σας εδώ. θα μας λείψει ο κύριος, με συγχωρείτε διορθώνει διερμένες, ο κύριος ο Σάλιβαν, γιατί ήταν πολύ συμπαθητικός και βέβαια εξαιρετικά ικανός, πάντοτε συνεργάστηκε μαζί μας όπου ήταν απαραίτητο. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να καταγράψουμε αυτή την επιστολή και να ευχαριστήσουμε επίσημα τον κύριο Σάλβαν για την πολύ θετική του συνεισφορά. για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο μας βοήθησε να προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε στο 4 και το σημείο 5 παράλληλα θα τα δούμε μαζί. Καταρχήν έχουμε την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την υποβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο 5 έχουμε την αντίστοιχη συμφωνία με τη Δημοκρατία του Καμερούν, ακριβώς για τα ίδια θέματα. Εμείς λοιπόν είμαστε η αρμόδια επιτροπή, η συγητής και στις δύο περιπτώσεις, και στις δύο περιπτώσεις είναι ο Γιάννικ Ζαντό των Πρασίνων. Να σας υπενθυμίσω μόνο πως το Δεκέμβριο του 2005 το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψει τέτοιου είδους εταιρικέ σχέσεις με τις χώρες παραγωγούς ξύλου στα πλαίσια των όσων αποφασίστηκαν το 2003 για την υποβολή, την υποβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλής για να αποφευχθεί το πρόβλημα της λαθρέας υλοτομίας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον Γιάννη Κζαντό για να μας τα πει με λεπτομέρειες. Με συγχωρείτε, έχουμε και ένα διαδικαστικό. Η Κάθρη νομίζω κάτι θέλει να πει. Όχι. Μετά τον Γιάννη Κζαντό θα της δώσω το λόγο. Γιάννη, μπορείς να προχωρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για δύο συμφωνίες εθελοντικές εταιρικέ σχέσεις. Είναι οι πρώτες που θα υπογραφούν, για τις οποίες γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο. Το 2009 υπεγράφει η σχετική εταιρική συμφωνία με την Κάνα, πριν όμως τη θέση εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνης. Είναι δύο φάκελοι αρκετά παρόμοιοι παρόλο που η πολιτική κατάσταση στο Κονγκό, Μπραζαβίλ και στο Καμερούν είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτό που θελήσαμε να λάβουμε υπόψη στο σχέδιό μας ε, ε, ε, στο θέμα του ότι ακόμα και η επίσημη υλοτομία μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ συνέπειες και αυτέ οι συμφωνίε εταιρική σχέση, επειδή ακριβώ καλύπτουν πάρα πολλέ από, αυτές τις, τα σημεία που μα ενδιαφέρουν είναι καλοδεχούμενε. Πρέπει να κάνουμε βέβαια μια διαφοροποίηση μεταξύ Καμερούν και Κονγκό αλλά και για τι δύο ε, περιπτώσει, θα γνωμοδοτήσουμε υπέρ τη επιβεβαίωση, τη έγκριση αυτή τη εθελοντική συμφωνία. Αντίθετα, έχουμε ένα αίτημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παρόλο που και στις δύο αυτές υποθέσεις οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων σεβάστηκαν μάλλον το πλαίσιο το οποίο έχουμε συμφωνήσει, σε επίπεδο διαβούλευσης ε, και διαπραγματεύσεων με την κοινωνία των πολιτών, νομίζω ότι νομιμοποιούμαστε να εκφράσουμε κάποιες ανησυχίες για τη θέση σε εφαρμογή αυτών των συμφωνιών εταιρική σχέσης. Γιατί θα σας το εξηγήσω. Αυτό που θα θέλαμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έξι μήνες έξι μήνες μετά τη θέση σε εφαρμογή των ε, συνθήκων αυτών, να μας παρουσιάσει σε μία έκθεση για τα μέτρα τα οποία όντως ελήφθησαν για να εφαρμόσουν τα όσα έχουμε συμπεριλάβει εμείς στις συμφωνίες. Και κυρίως στην περίπτωση του Κονγκό Μπραζαβίλ, η διαβούλευση και η συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών, πολιτών είναι μια δύσκολη ε, πτυχή. Για το Καμερούν τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Αυτό που θα θέλαμε είναι αρκετά σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει και να κινητοποιήσει και να πληροφορήσει εμάς για τους ειδικούς μηχανισμούς που θα χρησιμοποιηθούν για να εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες εταιρικέ σχέσης στα πλαίσια του, του ε, ευρύτερου προγράμματος FLECT. Να δούμε ποιοι είναι οι πόροι που είναι διαθέσιμοι, αν υπάρχει δυνατότητα τεχνικής βοήθειας, συνδρομής και πώς θα εφαρμοστούν αυτά. Και ένα συγκεκριμένο αίτημα που συνδέεται με το εξή υποθετικό σενάριο, δηλαδή το να είναι λυπής η εφαρμογή αυτών των ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης, είναι το να έχουμε κάποια διαιτησία την οποία θα μπορούσαν να ζητήσουν όλοι οι εταίροι που θα υπογράψουν αυτή την εταιρική σχέση Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα για τους πολίτες ε, του Κονγκό ή του Καμερούν με τη συμφωνία αυτή, νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει και ένας επιδιαιτητής, ο οποίος θα μπορούσε σε περίπτωση που η κυβέρνηση, για παράδειγμα, του Κονγκό ή της Καμερούν, του Καμερούν δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών, να αναλάβει το θέμα αυτό στα πλαίσια των ε, συμφωνιών, των θελοντικών συμφωνιών εταιρική σχέση. Ένα διαμεσολαβητή λοιπόν. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άγρυπνα να παρακολουθήσει την θέση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και να έρθει ενώπιόν μας για να μας εξηγήσει ακριβώς πού βρισκόμαστε γιατί ο στόχος των πρώτων αυτών συμφωνιών που περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να δημιουργήσουν προηγούμενο. Όχι μόνο για τα όσα έχουν ήδη λάβει χώρα. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν με πολύ σωστό τρόπο, αλλά για να δούμε επίσης και το θέμα της εφαρμογής. Να δώσω λοιπόν ε, στην Εύα Μπέρντε το λόγο πρώτη ηγήτρια. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως παραγωγοί και καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι κυβερνήσεις του Καμερούν και του Κονγκό έχουν υποχρέωση να εκριζώσουν την παράνομη ε, υλοτόμηση. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ενώ το συζητάμε εμείς αυτό το θέμα, οι συνάδελφοί μας ε, συνεδριάζουν στην Λαγκόγια, στην Ιαπωνία, σε μια προσπάθεια να φτάσουν σε μια συμφωνία για ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για την προστασία της βιοπικιλότητας. Ε, αυτό αποπειράται να δώσει οικονομική αξία στους φυσικούς φυσικούς πόρους. Η εκμετάλλευση και οι εξωτερικές βιομηχανίες, ιδιαίτερα οι ομάδες ε, υλοτόμηση που μέχρι στιγμής είναι τελείως απορριθμισμένη, οδήγησε στην ε, κρίζωση μεγάλων δασικών εκτάσεων στην Αφρική. Και τώρα υπάρχουν ε, πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι που στηρίζουν τις οικογένειές τους μέσω αυτής της υλοτόμησης. Λόγω έλλειψης ενημέρωσης αυτή η βιομηχανία έχει έχει διευκολύνει όχι μόνο την παράνομη και τελείω απορριθμισμένη υλοτόμηση, αλλά και την παράνομη εμπορική εκμετάλλευση της άγριας ζωής στην Κεντρική και Δυτική Αφρική. Ε, υπάρχει μεγάλη λοιπόν πίεση στους τοπικούς πληθυσμούς που ζουν στα δάση. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες όσον αφορά τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις της εμπορικής υλοτομίας στην άγρια ζωή. Οι Ευρωπαίοι και οι Αφρικανοί θα πρέπει να εστιάσουν στην ε, στήριξη των βιώσιμων πόρων και να δημιουργήσουν τι κατάλληλε πολιτικέ ώστε να προστατεύσουν τα δάση. Εγώ καλωσορίζω αυτή την ε, Συμφωνία εταιρική σχέση ω ένα εξαίρετο πρώτο βήμα, αλλά όπω ε, τόνισε και ο κ. Ζανό στην έκθεσή του θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και υπάρχουν ε, ερωτήματα σε σχέση με το γιατί η Ευρώπη χρησιμοποιεί τόσο πολύ τροπική ξυλία και σε σχέση με το πόσα πληρώνει για αυτή την ξυλία που φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ένα πολύ ακριβό προϊόν. Αυτά τα προϊόντα είναι όχι μόνο ζωτική σημασία σε οικότοποι για την άγρια ζωή, αλλά και πολύ σημαντικά για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Μόνο τα δάση του Καμερούν εκτιμάται ότι περιλαμβάνουν γύρω στις 30, ε, τα 30 δισεκατομμύρια φυτά κυβικά, δεσμεύουν 30 ε, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα άνθρακα ετησίω. ετησίως. Αυτά τα δάση ανήκουν σε ολόκληρη τη γη, παρότι είναι πόροι του ίδιου του Καμερούν. Είναι όμως ε, πόροι πολύτιμοι ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό και θα πρέπει να διατηρηθούν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτού του είδους τις συμφωνίες και θα πρέπει όντως να εφαρμοστούν και να επιβληθούν σωστά. Έχουμε καθήκον να στηρίξουμε τις καλές προθέσεις αυτών των χωρών και να τις βοηθήσουμε στη ε, διεθνή προγράμματα διαχείρισης ε, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτού του είδους της συμφωνίας, ε, στόχος των οποίων είναι πολύ θετικό. Και ιδιαίτερω καλωσορίζω την καινοτόμα διαδικασία μέσω της οποίας επετεύχθη η συμφωνία. Αυτή η νέα προσέγγιση στη διαχείριση των δασών, όπου δίνεται έμφαση στην κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή αυτής, έτσι ώστε οι πολιτικές καταρχήν να εγκρίνονται και μετά να, εφαρμόζονται και να αποτελούν αυτές την κανόνα. Αυτή η προσέγγιση θα είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία αυτή τη συμφωνία. Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση ακόμα μα περιμένει στη δύσκολη μετακίνηση από το κείμενο στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από του σκιώδεις εισηγητές. Ίσως κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο. Ο Τζο Χίγκιν από την ομάδα Γκουε. Χωρί μικρόφωνο ο κύριο Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο τους λαούς του Κονγκό και του Καμερούν, αλλά τους λαούς της Ευρώπης και ολόκληρη την Ιφίλιο. Νομίζω ότι ο Γιάννικ κάλυψε τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή μας και να τα λαμβάνει υπόψη, καθώς και να πιέσει όσον αφορά την εφαρμογή ετούτης της συμφωνίας και την επαλήθευση, την παρακολούθηση της εφαρμογής της. Προφανώς αν δούμε από κοινού το Καμερούν και το Κονγκό, και τις αιτήσει εξαγωγές τους εξηλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπουμε ότι είναι τεράστιες ποσότητες. Και το θέμα της ε, βιομηχανικής εκμετάλλευσης ε, μεγάλης κλίμακας των δασών οδηγεί στην αποδάσωση και την εξάλληψη πολλών ειδών. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλης ανησυχίας και εγώ στηρίζω έντονα το αίτημα του Ζανό ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εισάγουν την ξυλία από το Καμερούν και από το Κονγκό. Νομίζω πως είναι πραγματικά αποτροπιαστικό το να γίνεται καταστροφή δασών σε μεγάλη κλίμακα προς όφελος ιδιωτών στην ουσία. Ενώ πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πόρο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά και την βιοπικιλότητα. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν πολύ αυστηρέ ε, ρυθμίσεις ως προς αυτό. Και τώρα το να συνδεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιμείνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών από τις περιοχές από όπου προέρχεται η ξυλία είναι εξίσου σημαντικό. Είναι θέμα ζωής και θανάτου, ιδιαίτερα στο Κονγκό. Αν δει κανεί τι συμβαίνει εκεί με τον πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, ένα σωρό φρικαλαιότητες στις οποίες ε, υπόκειται ο τοπικός πληθυσμός εδώ και χρόνια. Το θέμα λοιπόν της παρακολούθησης των συμπεφωνημένων πρακτικών είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε όλη αυτή την υπόθεση. Πώς δηλαδή μπορούμε να γνωρίζουμε ότι γίνονται σεβαστά τα όρια, ότι γίνονται σεβαστές οι ποσοστώσεις, ότι δεν γίνονται χονδρική υλοτόμηση και εξαγωγή της ξυλίας. Τέλος, Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι... Ένα τομέα όπου η λογική χρήση των πόρων θα πρέπει να προηγείται των ιδιωτικών συμφερόντων των ε, ομίλων. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή από το είδος των ξύλων που έρχονται από το Κονγκό και το Καμερούν, που θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλο είδος ξυλία, ώστε αυτά τα τόσο σημαντικά δάση να διατηρηθούν και να μην καταστρέφονται με το ρυθμό που καταστρέφονται σήμερα. Και φυσικά οι απλοί άνθρωποι, οι πληθυσμοί του Καμερούν και του Κονγκό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η διατήρηση των δασών τους είναι προς όφελος, ολόκληρης, ανθρωπότητας, άρα λοιπόν η κοινωνία μας έχει ευθύνη να τους βοηθήσει ώστε να αναπτυχθούν όσον αφορά την απασχόληση, αλλά με τρόπο που να είναι βιώσιμος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν έχει να κάνει κάποια σχόλια. Στα όσα είπε ο εισηγητής και για τις προτάσεις του εισηγητή. Ποιος ε, αντιπροσωπεύει την Κομισιόν. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση ε, Ανάπτυξης και μαζί με κάποιους ακόμα συναδέλφους αρμόδιος για την πρόθεση αυτών των συμφωνιών. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαντό για την πολύ θετική αξιολόγηση που κάνει αυτών των εθελοντικών συμφωνιών εταιρική σχέση. Νομίζω ότι είναι πολύ καινοτόμε συμφωνίες, τουλάχιστον σε επίπεδο σύλληψης. Το είπε άλλωστε και η κυρία Μπίρντερ είναι κάτι το καινούριο σε διεθνές επίπεδο και το εντυπωσιακό είναι ότι σε διαπραγματευτικό επίπεδο ήταν τόσο ευρία η συμμετοχή και από τις δύο ενδιαφερόμενες ε, κυβερνήσεις. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Των Καταρχήν το ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση από πλευράς κυβερνήσεων είναι γνωστό. Το ενδιαφέρον είναι πως η κοινωτία των πολιτών αναλαμβάνει στις δύο αυτές περιπτώσεις το ρόλο του Μοχλού που θα ισορροπήσει την εσωτερική τάξη των πραγμάτων στο Καμερούν και στο Κόγκο γιατί Μόνο δημιουργώντας αυτού του είδους την ισορροπία μπορεί να επιβάλλουμε με αποτελεσματικό τρόπο την τήρηση αυτών των συμφωνιών. Τονίζω πως πρόκειται για θελοντικές συμφωνίες, δεν είναι δεσμευτικές. Οι κυβερνήσεις λοιπόν ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις σε θελοντική βάση και αφού λήξουν οι διαπραγματεύσεις αναλαμβάνει θελοντικά να σεβαστεί τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται, τους όρους και τις ρήτρε που εξασφαλίζουν πως οι συμφωνίες αυτές θα εφαρμοστούν και σύμφωνα με το πνεύμα και σύμφωνα με το γράμμα των όσων έχουν συμπεριληφθεί. Τώρα για την βιώσιμη διαχείριση των δασών άκουσα πολλά για την καταστροφή των δασών. Νομίζουμε πως οι συμφωνίες αυτές που βασίζονται στο εθνικό δίκαιο και που και στο Καμερούν και στο Κονγκό δημιουργούν τους κανόνες που θα οδηγήσει σε βιώσιμη διαχείριση των δασών. Θα βασιστούν πλήρως στην αρχή της βιωσιμότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή αυτών, γιατί μέσω αυτών των συμφωνιών έχουμε το, δημιουργούμε το πλαίσιο ε, το οποίο θα επιτρέψει και στους εθνικούς νόμους να γίνουν σεβαστοί. Γιατί επαναλαμβάνω το θέμα είναι η εφαρμογή και όχι η νομοθεσία τώρα για την αποψήλωση η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και ξεπερνάνε ε, τα όσα έχουμε εδώ στις συμφωνίες μας. Γίνονται πάρα πολλές, ε, πάρα συζητήσεις για το πώς μπορούμε να ανταμείψουμε τις χώρες που διατηρούν τα δάση σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέσα για να το επιτύχουμε. Θέλουμε λοιπόν μια διευρυμένη εντολή για την καταλληλότερη προστασία των δασών. Οι συμφωνίες αυτές μας δίνουν μια ευκαιρία να συζητήσουμε το νομικό πλαίσιο με τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και όπως ε, αναφέρει και η εισήγηση του κ. Ζαντό, το νομικό πλαίσιο υπάρχει και αποτελεί τη βάση από τις οποίες οικοδομήσαμε αυτές τις συμφωνίες. Έχουμε πολλά μέτρα συμπεριλάβει, για παράδειγμα έναν ε, έλεγχο που θα γίνεται σε αιτήσια βάση από ανεξάρτητο ε, ελεγκτή. Έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών, όπως επίσης και το δικαίωμα ένστασης και προσφυγής είτε προς τις οικίες κυβερνήσεις είτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε λοιπόν διάφορα μέτρα, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε στιγμή εκφραστούν ανησυχίες στο Κονγκό, στο Καμερούνι και σε κάποια από τις άλλες χώρες όπου θα υπογραφούν και στο μέλλον συμφωνίες πώς οι ανησυχίες αυτές θα μπορούν να εκφραστούν και να ακουστούν. Για έναν πιο αυστηρό μηχανισμό, τον οποίο θα πρέπει να σέβονται οι κυβερνήσεις, Ε, πιστεύω ότι αυτό θα ισχύσει και θα επιτρέψει να αναθεωρηθούν ε, την κατάλληλη στιγμή όλες οι διατάξεις που έχουμε συμφωνία. Τώρα για τις διάφορες κυβερνήσεις να σας πω ότι δεν μπορούν να κάνουν οι εθελοντικέ συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Δεν είναι το κατάλληλο μέσο αν θέλουμε να κάνουμε μία επισκόπηση του νομικού συστήματος που ισχύει σε κάποια συγκεκριμένη χώρα όπως λένε και οι Βρετανοί δεν είναι δυνατόν να αρχίσουμε από το τέλος για να φτάσουμε στην αρχή. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα πράγματα ανάποδα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να πιέσει και για να επιβάλλει συμφωνίες. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε όμως εδώ και την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση που μπορεί να προσφέρει. Δεν μπορεί όμως να αναλάβει εξ το ρόλο αυτό της επιβολής. Να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπεται μια ετήσια έκθεση πεπραγμένων εφαρμογής. Έχουμε μια μεικτή επιτροπή που θα παρακολουθεί σε διάφορα στάδια και σε τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή στις χώρες αυτές και οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να δώσουν ε, πλήρη δημοσιότητα στις εκθέσεις, όπως επίσης και στα όσα ε, θα ε, εμφανίζονται κατά τον ετήσιο έλεγχο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας υπενθυμίζω το προσωρινό χρονοδιάγραμμα που προβλέπει έγκριση της εκθέσεως στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου. Με συγχωρείτε, νομίζω θέλετε να σχολιάσετε. Εγώ θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Νομίζω πως υπάρχουν ένα-δύο σημεία επί των οποίων μπορούμε ακόμα να συζητήσουμε. Άκουσα όλα τα εργαλεία που υπάρχουν ήδη και πέρα από την ανεξάρτητη πυρογνωμοσύνη το θέμα της διαμεσολάβησης και του συστήματος ε, καταγγελιών είναι για μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή δεν απευθυνόμαστε μόνο σε κάποιον εξωτερικό σύμβουλο, είναι μια άλλη λογική. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε ανεξάρτητοι από τα συστήματα διακυβέρνησης των εν χωρών. Δηλαδή αυτές οι συμφωνίες ε, θέλουμε βέβαια να βοηθήσουν στην καλύτερη διακυβέρνηση των χωρών αυτών αν το μπορέσουν να το καταφέρουν τόσο το καλύτερο. Αλλά δεν μπορούμε να, εξαρτηθούμε, να εξαρτώμαστε μόνο από αυτές τις ε, κυβερνήσεις και δεν μπορούμε να αναμειχθούμε στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών. Ελπίζω πως θα έχουμε απαντήσεις αργότερα για τη διαφάνεια και για τη συνεργασία σίγουρα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε στο σημείο 6 εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου ζόρς Άμπεν Κούτας σε σχέση με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, με τις ΗΠΑ για τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την πρόθεση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν ειδικέ υποχρεώσεις σχετικά με υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 20 Δύο. ένα, με συγχωρείτε, της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, της ΓΚΑΤΣ. Ο κύριος Κούτας έχει το λόγο. Η γνωμοδότηση που ζητείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται αντισταθμιστικές αντισταθμίσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από αυτά που εξηγήσατε. Η αντιστάθμιση αυτή που είναι ένα πακέτο και που εγκρίθηκε αναφέρεται σε υποχρεώσεις, σε τεχνικές ε, υπηρεσίες και υπηρεσίες αποθήκευσης και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. Εγώ προσπάθησα να αναπτύξω μια συνενετική προσέγγιση συναντήθηκα με τις ε, πιο σημαντικές οργανώσεις του τομέα που με πληροφόρησαν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που ε, συμμετέχουν στον κλάδο έχουν σημειώσει ζημίες και μάλιστα έχουν κριθεί άδικα, αρνητικά από τις Αμερικανικές αρχές. Γι' αυτό και θα συστήσω στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις Αξιώσει και αιτήματα του τομέα για να εξασφαλίσει όσο γίνεται ίσως του ανταγωνισμού. Από την άλλη μεριά, η απόφαση των ΗΠΑ λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συμφωνίας Γκάτς και επομένως είναι απόλυτα νόμιμη. Η αντιστάθμιση που συμφωνήθηκε προέκυψε από συνεννοήσεις, από ε, ε, διαπραγματεύσεις επίσης νόμιμες αφού απορρέουν από, την, ε, από το ίδιο άρθρο οι κανόνες του ΠΟΕ αποδείχθηκε ότι είναι μηχανισμός επαρκής για να αποφευθούν εμπορικοί πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις. Τονίζω τέλος ότι πρόκειται για θετική συμφωνία, εγώ είμαι υπέρ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τις και τους συναδέλφους να υποστηρίξουν με την ψήφο τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ούρσουλα Χένικ. Όχι εσείς, καλά. Δεν επιθυμείτε να σχολιάσετε. Do you? So. <laughs> Okay. So no comment from the... Άρα δεν υπάρχει σχόλιο πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η διακόπτη ο γραμματέας, ο κ. Φιέλνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν ίσως να μην είναι διατεθειμένη ή έτοιμη να σχολιάσει αμέσω τώρα, αλλά ίσως αργότερα θα ήθελα να ζητήσω μια εξήγηση περί του τι είναι νέο σε αυτή την υπόθεση της αντιστάθμισης. Έχω ακούσει σχόλια από ενδιαφερόμενα μέρη που λέγουν ότι δεν προκύπτει τίποτε το νέο και ότι όλη η προσπάθεια απολύγει σε πράγματα τα οποία ήδη είχαμε και τέλο πάντων δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία σε σύγκριση με τις απώλειες του ε, τομέα των ε, τυχερών παιχνιδιών. Θα ήθελα λοιπόν από την Κομισιόν να ακούσω ποιο είναι το νέο στοιχείο σε σύγκριση με τα όσα είχαμε για παράδειγμα πριν ε, στον ταχυδροχυδρομικό τομέα, για παράδειγμα. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν κάτι σε κάποιο, σε κάποιο στάδιο. Μπορείτε να απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Όχι απαραίτητα τώρα. No, later. Κούτας. Uh, Εσείς κύριε Κούτας. Ευχαριστώ. Αν ε, δεν επιθυμεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πω στον συνάδελφό μου ότι εγώ συζήτησα με τις περισσότερες από τις ε, εταιρείε, τις μεγάλες τουλάχιστον, που εμπλέκονται στον τομέα. Και στράφηκε η συζήτηση γύρω από ένα απλό πράγμα. Κατανοούν τον θετικό χαρακτήρα της ε, συνένεσης αυτής, κατανοούν την θέση και τη δική μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και οι εταιρείε που έχουν σημειώσει ζημίες. Είπα ότι ορισμένες από αυτές έχουν υποστεί ζημίες. Ακόμα και αυτές λοιπόν συμφώνησαν ότι δεν είναι δυνατόν να προκύψει καλύτερη συμφωνία από αυτήν. Αυτό που ήθελαν είναι να αναγνωριστεί η κατάσταση αυτή και να γίνουν δεκτές. Να γίνουν Αυτό ζήτησαν από μένα ως Κύριε Φιέλεν, αν θέλετε να πιούμε ένα καφέ μαζί μετά για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Καταλαβαίνω πάντως αυτό που λέτε και επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόθεση από πλευρά Αμερικανού νομοθέτη να ανοίξει την αγορά στο τυχερό παίγνιο. Ίσως αργότερα να γίνει αυτό. Φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε λοιπόν κάποιες αλλαγές. Αλλά όχι για την ώρα. Άρα η αντιστάθμιση δεν θα πάει στον τομέα που έχει υποστεί τις ζημιές, αλλά αυτό που, είναι, που έχει κρίσιμη σημασία είναι το ερώτημα εάν υπάρχει κάποια ανάλογη ε, αντιστάθμιση για άλλους τομείς. Εγώ έχοντας μιλήσει σε διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν και διάφορους εμπειρογνώμονες, έχω την αίσθηση ότι τις μέρες από τις αντισταθμίσεις που έκανα και ιδίως στα ταχυδρομεία, αντισταθμίζουν κάπως την ε, ζημιά του τομέα των τυχαίων παιχνιδιών. Στο σύνολο δηλαδή το γεγονός ότι απέσυραν τις δεσμεύσεις τους σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρουν ε, αντίστοιχη πρόσβαση στην αγορά κάπου αλλού. Για να μπορέσω λοιπόν να κρίνω εγώ, ίσως να είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να επιτύχουμε, αλλά θέλω να μάθω αν υπάρχει κάποια ισότητα, αν υπάρχει κάποια κάποιο χαρακτήρα δίκαιο, α πούμε, ή μήπω απλώ μας περιπέζουν οι ΗΠΑ λέγοντας ότι αποσύρουμε αυτό το μεγάλο τομέα και σας δίνουμε ένα μικρό ε, σε αντιστάθμιση. Ε, ίσως να είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε, αλλά τουλάχιστον να διαμαρτυρηθούμε έντονα. Α, τον υπολογισμό θα ήθελα να έχω, δεν τον έχω μάθει ακόμη και θα ήθελα να τον έχω στα χέρια μου πριν να ψηφίσω. Έχετε ε, κάποιο ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο δεν είστε διατεθειμένοι να απαντήσετε, κυρία Χένιχ. Ορίστε. Μάλλον επειδή δεν πρόλαβα να σηκώσω το χέρι μου. Ε, βέβαια υπάρχει κάτι το νέο. Οι δεσμεύσει αυτές είναι νέες και εμείς προτείναμε την συμφωνία αυτή για απόφαση του Συμβουλίου διότι ε, θεωρούμε ότι είναι καλή η συμφωνία γι' αυτό και την συνάψαμε. Τώρα ταχυδρομικές υπηρεσίες και τα λοιπά, ε, χώροι αποθήκευσης, τεχνικές υπηρεσίες και ορισμένες άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεως είναι πλήρης δεσμεύσης, δηλαδή αναλαμβάνει πλήρως τη δέσμευση η άλλη πλευρά των ΗΠΑ και εγγράφονται πλέον αυτές στο χρονοδιάγραμμά τους. Μπορεί κανείς να εξετάσει εάν θα αλλάξει αυτό το πράγμα την κατάσταση στην αγορά, αλλά οι δεσμεύσεις αυτές συχνά είναι, έχουν δεσμευτική ισχύ, νομική δεσμευτική ισχύ για την αγορά. Αυτό μπορεί να κάνει κανείς. Αλλά πάντως αυτές είναι νέες δεσμεύσεις εξορισμού και εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστή έκβαση διαπραγματεύσεων που είχαν δύσκολο χαρακτήρα. Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή για την ολοκλήρωση της συζητήσεως, το λόγο με έχει ζητήσει ο κ. Ιακολίνο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα την χαρά να ακούσω την πλήρη παρέμβαση του εισηγητή, αλλά άκουσα τον προηγούμενο συνάδελφο από το ΕΛΚ και της Κομισιόν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ίσως κάτι πιο συγκεκριμένο στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών προσαρμογών θα έπρεπε να καθοριστεί. Το να μιλάμε έτσι γενικά χωρίς συγκεκριμένη διευκρίνηση των μέτρων αυτών, του βαθμού αυτών των προσαρμογών δεν είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος το είχαμε ζητήσει νομίζω και ολοκληρώνω με αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Είχαμε ζητήσει από τον εισηγητή Κούτας να προσθέσει στην παρέμβαση, την οποία εγώ κατέγραψα ε, ευνοϊκά, να μας δώσει και ένα προφίλ για την υγειονομική προστασία των ε, εργαζομένων εκεί, ειδικά όταν αυτοί ε, μείβονται. Και πόσα αμείβονται. Ο Μπαρνιέ ξεκίνησε πρόσφατα με μεγαλύτερη σαφήνεια από ό,τι, από στο παρελθόν ένα πράσινο βιβλίο για τα τυχερά παιχνίδια online. Ευχαριστώ. Κύριε Κούτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους που, που παρενέβησαν. Φυσικά, πείτε μου τι θέλετε να βελτιώσουμε στην έκθεση, αλλά μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μια συνένεση, μπορούμε να πούμε ναι ή όχι. Ίσως στις επεξηγηματικές σημειώσεις να προσθέσουμε κάτι, να αφαιρέσουμε κάτι, αλλά μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είμαι φυσικά ανοιχτός να συζητήσουμε, αν έχετε ε, ιδέες μπορούμε να τις συζητήσουμε μεταξύ μας και να μην ε, τρώμε το χρόνο της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Για την υποβολή τροπολογιών έχουμε προθεσμία 29 του μηνός και μην ξεχνάτε, επειδή πρόκειται για φάκελο συνένεσης, μόνο ένα είδος τροπολογίας είναι δυνατό, δηλαδή μια τροπολογία που προτείνει αντίθετη θέση από αυτή του εισηγητή. Προγραμματισμένη ημερομηνία για ψηφοφορία στην Επιτροπή είναι η 1η Δεκεμβρίου 2010 με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα μας έχει, θα έχει έρθει σε επαφή μαζί μας το Συμβούλιο για αυτό το θέμα, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί μας. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 7. Είναι μια παρουσίαση της Επιτροπής. Η πρόταση εδώ είναι λοιπόν πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν. Υπευλήθη στο Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας παρουσιάσει το θέμα. Ξέρετε ότι μετά τις ε, τρομερές πλημμύρες στο Πακιστάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κάποια μέτρα που θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόταση κανονισμό έτσι ώστε μόνο μερός να ανασταλούν κάποιοι δασμοί εισαγωγικοί από το Πακιστάν για, τρεις χρόνες, για τρία χρόνια. Είναι κυρίως υφαντουργικά, υφαντουργικά προϊόντα, 75 σειρές προϊόντων, δηλαδή 900 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό 27% λοιπόν των ε, ε, εισαγών από το Πακιστάν θα απαλλαγούν. Μιλάμε λοιπόν για μία αύξηση εισαγωγών από τη χώρα αυτή της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2009 με μια παράλληλη μείωση των εσόδων από τους ε, εισαγωγικούς δασμούς των 380 εκατομμυρίων ευρώ. Μια και μιλάμε για ε, μια ε, μοναδική τέτοια περίπτωση χορήγησης εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν, θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει την άδεια του ΠΟΕ στη Γενέβη. την ευκαιρία να συμμετάσχω σε διμερείς που έγιναν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, όπου συζητήσαμε μόνο εμπορικά θέματα και ένα από αυτά ήταν ο προτινόμενος κανονισμός. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στη χώρα του αυτό ο κανονισμός και ζήτησε να εγκριθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να διαβεβαιώσω τον Υπουργό πώς κατά την άποψή μου θα πρέπει να στηρίξουμε το Πακιστάν σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύει και νομίζω πως η Επιτροπή μας έχει την υποχρέωση να, να εξετάσει κατά πόσο επιβαρύνει υπερβολικά τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία ολόκληρο τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός αυτός. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο για να μας πει κάποιες ε, παραπάνω λεπτομέρειες για τον κανονισμό αυτό. Ο Ιγνάσιο Γκαρσία θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ και να σας παρουσιάσω επίσημα στην Επιτροπή σας αυτό το σχέδιο κανονισμού, παρόλο που είχαμε την ε, ευκαιρία και κλεισμένο των θυρών να συζητήσουμε το θέμα πριν από μερικές εβδομάδες. Ξέρετε πως ε, η πρόταση αυτή ακολούθησε μια ομόφωνη, ένα ομόφωνο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να προσφέρουμε συνδρομή στη χώρα αυτή στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει, όχι μόνο να προσφέρουμε λοιπόν ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να παρουσιάσουμε και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εμπορικών μέτρων. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήθηκε να καταθέσει προτάσεις τον Οκτώβριο, αυτό κάναμε, και μας ζητήθηκε να λάβουμε υπόψη την ε, βιομηχανική ευαισθησία για θέματα αυτά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τώρα, στην παρουσίαση που κάνω, να εξηγήσω κάποια από τα θέματα τα οποία θίξατε και εσείς και τα οποία ενδεχομένως να ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας, την Επιτροπή σας με συγχωρείτε, και βεβαίως θα απαντήσω και σε όποιο συγκεκριμένο θέμα θέλετε να θέσετε. Και βέβαια μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, ένα διάλογο αφού αποφασίζετε εσείς ποιος θα διοριθεί εισηγητής. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω ιδιαίτερα καταρχήν ποιος θα είναι ο κατάλογος προϊόντων που έχει συναυθεί σε αυτή την πρόταση κανονισμού έχει επιλεγεί, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία η πρόταση και τέλος δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, για τον κατάλογο προϊόντων που καλύπτει η πρόταση κανονισμού. Αυτό που θεωρήσαμε σημαντικό είναι να εξετάσουμε με πολύ συστηματικό τρόπο και με πολύ μεθοδικό τρόπο ποια είναι τα προϊόντα που θα απαλλάξουμε. Είπαμε λοιπόν πως οποιοδήποτε προϊόν το οποίο εξάγεται από το Πακιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο υπόκειται σε εξαγωγικούς δασμούς εφόσον γίνεται η εξαγωγή σε ελάχιστες ποσότητες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια αυτής της πρότασης εξαίρεσης. Αυτό λοιπόν ήταν το σημείο αφετηρίας. Όλα λοιπόν τα προϊόντα τα οποία δεν είναι ε, κλωστοϊφαντοργικά συμπεριλήφθηκαν στην πρότασή μας με δύο εξαιρέσεις. Το ρύζι που είναι πολύ βασικό τρόφιμο και θεωρήσαμε πως δεν είναι κατάλληλο να τοποθετηθεί στην πρότασή μας. Και το άλλο στο οποίο επιβάλλονται δασμοί, ένα άλλο ε, ε, προϊόν, στο οποίο επιβάλλονται κάποια αντισταθμητικοί δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Πακιστάν σε έστω και ελάχιστε ποσότητε θα απαλλαγούν. Δεύτερον, είμαστε πολύ ενημερωμένοι για την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζουμε τον ε, κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας στην Ευρώπη και γι' αυτό δεν έχουμε συμπεριλάβει 47 σειρέ προϊόντων ή ενδυμάτων που εξάγει στις χώρες μας το Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν απλώς τα σεντόνια, ε, τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητο προϊόν και έχει και κάποιο, ε, εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. 47 ε, λοιπόν είναι τα προϊόντα τα οποία αποκλείσαμε. Δεύτερον, εθανόλη. Είναι ένα προϊόν το οποίο και αυτό είναι ευαίσθητο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είπαμε θα το συμπεριλάβουμε αλλά θα δώσουμε ε, ε, τελωνιακό κωδικό. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε να είμαστε ε, σίγουροι πως ε, το βάρος αυτής της ε, πρότασης θα μοιραστεί ισότιμα και δεύτερον γιατί για τον οικονομικό αντίκτυπο εσείς μιλήσατε για 100 εκατομμύρια τα οποία υπολογίζουμε εμείς πως θα είναι η αύξηση των εισαγωγών που θα προκύψει από την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα έπρεπε να αναφερθώ σε κάποια επιπλέον στοιχεία για να σας εξηγήσω τι λάβαμε υπόψη. Συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή των προϊόντων τα οποία καλύπτονται από την πρότασή μας είναι 24 δις ευρώ. Αν λοιπόν κάνουμε μία σύγκριση θα διαπιστώσουμε πως η επίπτωση είναι μικρότερη από το 0,5% της ε, παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικές εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το αίτημα απαλλαγής είναι 15 δις. Αυτό και πάλι σας δίνει μια αίσθηση της σχετικής ε, σημασίας και σοβαρότητας των όσων προτείνονται. Όπως επίσης και του δημοσιονομικού, της δημοσιονομικής επίπτωσης. Θεωρούμε λοιπόν πως αυτό χρειάστηκε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε πως η πρόταση που σας καταθέτουμε είναι φιλόδοξη και θα δώσει επιπλέον ε, δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά στο Πακιστάν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και που παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν αρκετά προϊόντα ένδυσης και κλωστεφαντουργά δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση αυτή. Τώρα, για τα κράτη-μέλη και το πώς θα επηρεαστούν νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο γιατί η οικονομική συγκυρία ε, και το γεγονός πως τα βαμβακερά είναι πολύ ανταγωνιστικό το Πακιστάν είναι δεδομένο πως θα το αισθανθούν περισσότερο τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν βαμβακοβιομηχανία. Αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο της οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε και επαναλαμβάνω ε, συνολικά η επίπτωση είναι σχετικά μικρή. Χρονοδιάγραμμα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζουμε πως είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε την, ε, να πλαισιώσουμε μάλλον αυτή την απόφαση που ήταν ε, λήφθη ομόφωνα ε, με μία πρόταση που ανοίγει εξαγωγικές ευκαιρίες για το Πακιστάν. Ελπίζουμε λοιπόν να εγκριθεί η απαλλαγή στη Γενέβη πριν τα τέλη της χρονιάς. Στόχος μας είναι να υποβάλουμε το αίτημα εξαίρεσης μέχρι τις 11 Νοεμβρίου για να εγκριθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς και ελπίζουμε πως αυτό θα συνοδευτεί και από μια σχέση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβόλιο που θα επιτρέψει έγκριση του κανονισμού και πάλι μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Εμείς είμαστε σίγουροι πως θα πρέπει να δράσουμε στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ. Είναι λοιπόν ένας κανονισμός που θα εφαρμοστεί μόνο αφού χορηγηθεί αυτή η απαλλαγή στη Γενέβη, σύμφωνα επαναλαμβάνω με τα όσα διατάσσει ο ΠΟΕ. Αυτά ήθελα να ξεκαθαρίσω. Είμαι σίγουρος πως θα ακούσουμε πολλές ερωτήσεις για τα διάφορα στοιχεία της πρότασης και με μεγάλη χαρά θα απαντήσω. Βεβαίως Αφού οριστούν οι εισηγητές θα χαρώ πολύ να συναντηθώ μαζί τους και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και να δώσω πιο λεπτομέρειες απαντήσεις για οποιαδήποτε θέματα προκύψουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρώτη παρουσίαση, το οποίο, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη. Προσωπικά εγώ ζήτησα από το τμήμα πολιτικής στο Policy Department ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει μια μελέτη επιπτώσεων για τα μέτρα αυτά. Και έχω απευθύνθει και στον Επίτροπο κύριο Ντεγκούχτ μία σειρά ερωτήματα τα οποία εδώ δημόσια θέλω και πάλι να εκφράσω πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο ε, να έχουμε αυτή την τριετή διάρκεια. Μιλάμε για μια ε, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άρα λοιπόν δικαιολογούνται τα τρία έτη. Εμπορικές προτιμήσεις τριών ετών έκτακτης ανάγκης. Δεύτερον, δεν μπορώ να σας πω πως ε, τα όσα είπατε για την εθανόλη ε, μου εξήγησαν το θέμα. Γιατί, με συγχωρείτε, γιατί βρίσκεται την εθανόλη πιο ευαίσθητοι από άλλα προϊόντα, για παράδειγμα κλωστιφαντουργικά... και οι κλωστιφαντουργικές ε, εισαγωγές είναι ενδεχομένως εξίσου ευαίσθηση και περισσότερο ευαίσθητες, ευαίσθητο θέμα ε, στα, σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εκτός εάν θεωρούμε πως κάποια κράτη είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα όταν συζητάμε το θέμα των εμπορικών προτιμήσεων που χορηγούνται σε τρίτες χώρες και έτσι προκύπτει και η αθανόλη. Τρίτον, με εντυπωσίασε το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε τις πληροφορίες ε, επί των οποίων επιλέγησαν αυτά τα προϊόντα και λήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η Επιτροπή η δική μας του Κοινοβουλίου μπορεί να συζητήσει το θέμα χωρίς να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα έχει τέτοια στοιχεία στα χέρια της. Στοιχεία που να έχουν οδηγήσει στην επιλογή των εμπορευμάτων που έχουμε ε, στον κατάλογο. Ποσοστώσεις για κάποιες εισαγωγές ε, κατάρριξη ποσοστώσεων, για κάποιες άλλε νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας παράξει αυτές τις πληροφορίες. Τέταρτον, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λέει τίποτα για οποιαδήποτε ρήτρα εξασφάλισης, διασφάλισης για καταστρατήγηση των κανόνων και την εισαγωγή άλλων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατανοεί πως τα τρία έτη είναι υπερβολικά πολλά και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους μηχανισμό ασφαλείας που να μας εξασφαλίζει πως οποιαδήποτε αρνητική δυσάρεστη έκπληξη να αποφευθεί. Γιατί να μην έχουμε, να μην γίνει μια αναθεώρηση για παράδειγμα στο τέλος του της εκπνοής του πρώτου έτους, ε, να δούμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις και οι συνέπειες, να αξιολογηθούν αυτές και ενδεχομένω, εάν δούμε ότι είναι πολλές αρνητικές επιπτώσεις, να αναστείλουμε κάποιες από τις απαλλαγές. Εμείς θα προσφέρουμε στο Πακιστάν μία πολύ σημαντική εμπορική προτίμηση χωρίς να λάβουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε τουλάχιστον από το Πακιστάν να εγκαταλείψει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα νήματα, τα βαβακερά νήματα για παράδειγμα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ελαφρύνει τις αρνητικές συνέπειες από αυτές τις επαλλαγές που θα προσφέρουμε εμείς για κάποια κράτη και κλάδους. Βεβαίω και πρέπει να ζητήσουμε αυτή την ε, απαλλαγή από τον ΠΟΕ. Να εγκριθεί και εκεί. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά φαντάζομαι πως και αρκετά κράτη εκεί δεν θα ικανοποιηθούν ιδιαίτερα από το γεγονός πως προσφέρουμε αυτές τις εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν, γιατί θα επηρεαστούν. Γιατί βέβαια τμήμα των δικών τους εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί. Δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν χρειάζεται άλλωστε να αναφέρω ονόματα κρατών. Αναρωτιέμαι όμως Εάν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει σκοπό να τους εξαγοράσει μέσω κάποιων άλλων εμπορικών προτιμήσεων για να δεχτούν να χορηγήσουν αυτή την απαλλαγή. Αυτό έχετε σκοπό να κάνετε. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσει στη Γενέβη δυσκολίες. Πώς θα το αντιμετωπίσει. Με κάποιες παραχωρήσεις, για παράδειγμα, στη Βραζιλία για την Εθανόλη. Γι' αυτό λοιπόν δόθηκε ποσόστοση στην εθανόλη. Δίνω το λόγο συναδέλφους. Thank you very much. κύριος Φιέλνερ, ευχαριστώ. Θα αρχίσω με λίγο διαφορετικό τρόπο, ε, αντίθετα από σας κύριε Πρόεδρε. Το συζητήσαμε το θέμα στο Στρασβούργο και ήδη εγώ τότε είπα ότι με ικανοποιεί η πρόταση της Επιτροπής. την οποία βρίσκω λογική και ότι προσφέρει ένα καλό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η γνωστή καταστροφή στο Πακιστάν. Μάλιστα με εντυπωσιάζει και το Συμβούλιο που μπόρεσε να εγκρίνει τόσο γρήγορα. Νομίζω ότι πρέπει στη σημερινή εποχή να συνδυάσουμε τη βοήθεια με το εμπόριο. Τι νόημα έχει το να προσπαθούμε να βοηθήσουμε μια χώρα αν παρόλα αυτά της επιβάλλουμε δασμούς και έτσι κάνουμε πιο δύσκολο για την συγκεκριμένη χώρα που χρειάζεται βοήθεια να προβαίνει σε εξαγωγές. Λοιπόν νομίζω ότι είναι μια σύγχρονη στάση να συνδυάζουμε aid και trade. Και επίσης το γεγονό ότι ε, παρήχθη τόσο γρήγορα η απόφαση αυτή, η πρόταση αυτή, είναι σωστό. Εγώ θα έλεγα μάλλον ότι είναι καλή, αλλά δεν είναι επαρκή. Αυτή θα ήταν η συνήθι μου αντίδραση. Αλλά ε, έχοντα ακούσει τι συζητήσει. και τις κριτικές με τις οποίες δεν συμφωνώ, αλλά ε, βλέπω με ποια λογική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε αυτές τις 47 ε, γραμμές. Εγώ ο ίδιος δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Θα έλεγα όσο το δυνατόν περισσότερες. Αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες και εν και της κριτικής που ασκήθηκε από διαφόρους συναδέλφους και από συγκεκριμένες χώρες μέλη βέβαια και καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο έκανε όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένας τομέας όπου διαρωτώ με γιατί, για την εθανόλη δηλαδή. Θα έλεγα το ίδιο όπως ο πρόεδρος, αλλά με τον αντίστροφο τρόπο. Γιατί την εθανόλη. Ε, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου προοπτική ποτέ δεν κατανόησα γιατί πρέπει να επιβάλλονται δασμοί στην ενέργεια. Ειδικά όταν μιλούμε και για ασφάλεια των προμηθειών ενέργειας και πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και μάλιστα βιοενέργεια, οργανική ε, ενέργεια. Λοιπόν, υπό τις συνθήκες αυτές, εάν μπορούμε να μειώσουμε, να καταργήσουμε τους δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις για κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και μιλούμε εκεί επί ώρες και ώρες για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ενέργεια από βιολογικούς πόρους στην Ευρώπη. Και λοιπόν για ενέργεια τέτοια προέρχεται από το Πακιστάν και που γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε δεν καταλαβαίνω καθόλου. Ίσως είναι ευαισθησία κάποιων κρατών μελών. Αλλά από μια συνολική επισκόπηση του συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι είναι καλύτερα να μην υπάρχουν δασμοί. Πάντα είναι δύσκολο να δείξει κανείς αλληλεγγύη, αν και μιλούμε πολύ εδώ για αλληλεγγύη στην Ευρωβουλή. Όταν όμως καλούμαστε να ψηφίσουμε υπέρ της τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Διότι μεταξύ άλλων όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες στη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου υπέρ της οποίας θα δείξουμε αλληλεγγύη τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ψηφίσουμε. Πιο πολύ αλληλεγγύη με την υφαντουργία στην Ευρώπη με τα θύματα της, ε, των πλημμυρών στο, στο Πακιστάν. Ελπίζω πάντως η Ευρωβουλή να δείξει το ίδιο θάρρος όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Καταλαβαίνω βέβαια ποιε είναι οι συνέπειε, οι επιπτώσει όλων αυτών, αλλά μην λησμονούμε ότι πρόκειται για εξαιρετικέ συνθήκε και επομένω εξαιρετική πρόταση. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, όπω λένε μερικοί, ναι μεν εξαιρετικά μέτρα, αλλά με εξαιρέσει εξαιρέσεων. Αυτό για μένα δεν είναι πλέον κατανοητό. Μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να δώσει να ανοίξει περισσότερο το εμπόριο. Δίνουμε εμπορικές προτιμήσεις επειδή ελπίζουμε ότι θα αυξήσουν το εμπόριο με την Ευρώπη. Γιατί αν δεν μιλούμε γι' αυτό, αν δεν μιλούμε για αύξηση των εξαγωγών τους προς την Ευρώπη, δεν καταλαβαίνω καν γιατί μιλούμε τότε. Εάν μια τέτοια πρόταση δεν πρόκειται να έχει απολύτω καμία επίπτωση στι εξαγωγέ προ την Ευρώπη, δεν έχει και νόημα να γίνει. Ελπίζω πράγματι το Πακιστάν να αυξήσει τι εξαγωγέ του προ την Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η βασική ιδέα ε, της προσπάθειας αυτής δηλαδή να ενισχυθεί η ανάπτυξη της χώρας τους μέσω του εμπορίου. Εγώ δεν θα έλεγα ότι μία τριετία είναι μακρό ε, χρονικό διάστημα. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι είναι πολύ βραχή. Θα ήθελα μάλιστα όπως και ο πρόεδρος να ακούσω για ποιο λόγο επιλέχθηκαν τα τρία χρόνια. Και πάλι όμως εδώ θα το έβλεπα από την άλλη πλευρά. Γιατί τρία χρόνια και όχι πέντε. Και τέλος θα ήθελα να μάθω τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάλι όπως ο Πρόεδρος, πώς θα αντιμετωπιστεί, πώς θα το δεχτεί αυτό, ε, αυτή την πρόταση ο ΠΟΕ. Θα αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις εκεί. Ε, τι αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. με την πρότασή μας αυτή για να προσφέρουμε τη δυνατότητα στο Πακιστάν να επανέλθει και να αυξήσει την ευημερία ε, των κατοίκων του μετά με μια ανάπτυξη της οικονομίας. Ευχαριστώ. Ζαντώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν για την τριετή περίοδο. Το θέμα αφορά λιγότερο το ενεκλωστό υφαντουργία και περισσότερο την εθανόλη. Γιατί αυτό είναι και η ουσία του πακέτου αυτού για το Πακιστάν. Ποιον θέλουμε να βοηθήσουμε μέσω αυτού του επίγοντος πακέτου. Θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιες επιχειρήσεις ή το λαό του Πακιστάν. Α, στην αρχή είχα την εντύπωση πως η εντολή που έδωσε το Συμβούλιο και η Κομισιόν ήταν να διτυπώσουν μια πρόταση που θα επέτρεπαν να βοηθηθεί ο πληθυσμός του Πακιστάν. Όμως, όπως το γνωρίζετε, η ζάχαρη είναι ένα αγαθό εξαιρετικά πολύτιμο, είναι ένα σημαντικό τρόφιμο, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα πληθυσμό που ε, υποφέρει από τροφική ανασφάλεια. Και όταν βλέπουμε την κατάσταση ζάχαρη στο Πακιστάν ε, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε όπως και στον κόσμο ότι η μετατροπή σε καλλιέργειες για τα καύσιμα, τα βιοκαύσιμα ε, γίνεται εις βάρος της παραγωγής ε, ζάχαρης πολύ συχνά. Άρα το ερώτημα είναι σχετικά απλό. Πώς η Κομισιόν με την εντολή της ενίσχυσης ή βοήθειας ε, του πακιστανικού λαού για να αντιμετωπίσει την ανασφάλεια, την τροφική προβλέπει αυτή την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών εθανόλης προς την Ευρώπη. Δεύτερη ερώτηση, ποια είναι η ανάλυση που προβλέπει η Κομισιόν όσον αφορά την εξέλιξη της αγοράς της ζάχαρης στην ιστορική αγορά του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια για να ενσωματώσει τις επιπτώσεις της αύξησης της τοπικής παραγωγής ζάχαρης σε σχέση με την ε, εθανόλη. Τρίτη παρατήρηση, ποιες είναι οι γνώσεις της Κομισιόν όσον αφορά τις συνθήκες ε, καλλιέργειας της ζάχαρης στο Πακιστάν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι προβληματίζουν ε, τα θεσμικά όργανα η βιωσιμότητα των ε, βιοκαυσίμων. Και τελευταία ερώτηση που έχει περισσότερο νομικό χαρακτήρα, πώς η Κομισιόν θα εξετάσει την προέλευση της ζάχαρης. Το Πακιστάν έχει θέσει σαν στόχο την επάρκεια σε ζάχαρη δεν το έχουν ακόμα καταφέρει. Ένα κομμάτι της ζάχαρης, ένα τμήμα ζάχαρης ε, εισάγεται. Πώς λοιπόν η Κομισιόν προβλέπει την αύξηση της ποσόστοσης εξαγωγών βιοκαυσίμων από το Πακιστάν σε σχέση με την ίδια την προέλευση της ζάχαρης. Θεωρεί ότι αυτό θα ανταποκριθεί στο άρθρο 1 για τις εμπορικές προτιμήσεις που αφορά ζάχαρη πακιστανικής προέλευσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. David Camper. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε την εξής κατάσταση στο Πακιστάν. Έχει το Πακιστάν πυρηνικά όπλα ε, έχει ε, σχέσεις πιθανότατα με την ε, Αλ-Κάιντα, με προβλήματα βόρεια με τους Ταλιμπάν. Πρόσφατα επλήγει από φοβερές πλημμύρες και βλέπουμε μία πρόταση τώρα εδώ που σε 47 διαφορετικούς τομείς δασμών καταργεί τους κρατικούς δασμούς. Εδώ έχω ένα κείμενο Πραγματικά έχουμε ένα ευκολόγιο φραγμών, ποσοστώσεων, δασμών και πραγματικά διαρωτάμε. Έχει νόημα να βάζουμε τα συμφέροντα, τα προστατευτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από τη ε, θέματα ασφάλειας. Δηλαδή σπρώχνουμε στην ουσία το Πακιστάν στα χέρια των εξτρεμιστών. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον όσων κάθονται εδώ σε αυτή την αίθουσα, ούτε και αυτών που βρίσκονται εκτός της αιθούσης. Ευχαριστώ. Ο Τζο Χίγγινς, Γκούε. Πρόεδρε, Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι με κάποια λογική στην Ευρώπη, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού, θα συμφωνούσε ολόψυχα με την ανάγκη να βοηθηθούν οι άνθρωποι του Πακιστάν που υποφέρουν. Όταν έχουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν σοβαρά πληγή από τις πλημμύρες και την κρίση είναι τέσσερις φορές ο πληθυσμός της Δημοκρατίας της ε, Ιρλανδίας. Δηλαδή είναι μια τεράστια καταστροφή, όπως και αν τη μετρήσει κανείς. Όμως και εγώ θέλω να απευθύνω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα στον κύριο Γκαρσία της Επιτροπής. Γιατί το Συμβούλιο περιορίστηκε σε αυτό το στενό τρόπο προσπαθώντας να βοηθήσει τον λαό του Πακιστάν να ξεπεράσει την καταστροφή και η Κομισιόν έχει προβεί σε ανάλυση του ποιος πραγματικά θα ωφεληθεί κατά τη διάρκεια την τριετή αυτών των προνομίων. Αυτοί που υποφέρουν στο Πακιστάν είναι οι φτωχότεροι των φτωχών, είναι οι γεωργοί στα μικρά αγροκτήματα και οι εργαζόμενοι. πώς θα επηρεάσει η πρόταση αυτή τις ζωές τους προς το καλύτερο. Και πώς γνωρίζουμε πώς δεν θα ωφεληθούν περισσότερο οι πακιστανοί καπιταλιστές χωρίς να δώσουν κανένα επιπλέον εισόδημα σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Σε μια χώρα που είναι ιδιαίτερα κακόφημη όσον αφορά την διαφθορά που επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες. Πώς ξέρουμε πώς δεν θα ωφεληθούν από αυτά όλα οι διεφθαρμένοι δημόσιοι πάλι. Τι κάνετε ως προς αυτό. Και Πρόεδρε, ένα από τα θέματα κλειδί για στο Πακιστάν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα των τροφίμων, της επιβίωσης των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά, για παράδειγμα, χρειάζονται περισσότερη τρόφιμα και ασφάλεια στα τρόφιμα. Υπάρχει δηλαδή επιστημιστική κρίση. Και αυτό επηρεάζεται και από τις φεουδαρχικές ε, καταστάσεις που επικρατούν ακόμα στο Πακιστάν. Υπάρχει ένας ε, φεουδάρχης όπως υπήρχε το 19ο αιώνα στην Ιρλανδία με τεράστιο κόστος για τον απλό λαό. Γιατί λοιπόν δεν έχετε λάβει υπόψη ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε στην παραγωγή, μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, ας πούμε με την παροχή σπόρων ή ε, βιώσιμων λιπασμάτων και να παρασταθούμε στον τοπικό πληθυσμό για την παραγωγή τροφίμων. Το ήταν αυτό ένα θέμα κλειδί. Όπως ε, και ολόκληρη αυτή η ιδέα λόγω της, ε, των αναγκών στο Πακιστάν, στο Πακιστάν γίνεται τεράστια κερδοσκοπία στις ε, παγκόσμιες αγορές τροφίμων, ενώ ο κόσμος λιμοκτονεί στη χώρα αυτή. Είναι πραγματικά διαστική κατάσταση. Και επίσης, Πρόεδρε, προς την Επιτροπή απευθύνομαι. Έχετε εξετάσει πώς η αποπληρωμή των χρεών επηρεάζει τον λαό του Πακιστάν οι πόροι που θα μπορούσαν να στραφούν στην ανακούφιση των όσων υποφέρουν από κακή διατροφή ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση των εκατοντάδων σπιτιών που έχουν καταστραφεί. Ε, σκεφτήκατε την ακύρωση χρέους, ώστε να μπορέσουν να διοχετευθούν πόροι προς αυτές τις κατευθύνσεις. Εγώ νομίζω πως είναι μια πολύ στενόμυαλη πρόταση Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Θα δώσω και πάλι το λόγο στην Επιτροπή και να διευκρινίσω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά του να βοηθηθεί το Πακιστάν μέσω του εμπορίου. Ε, θέλω όμως να μου διευκρινίσετε αυτή την ασυνέπεια που υπάρχει μέσα στην πρόταση της Κομισιόν και δεύτερον, ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Γιατί όταν σκεφτούμε την ε, αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς το Πακιστάν, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι από τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης, μόνο 6-7 θα πληρώσουν. Αυτή είναι η ερώτησή μου, ο Κρίστοφερ Φιέλνερ. Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Αλλά πιστεύω πως ολόκληρη η ιδέα του να χρησιμοποιηθεί το εγώ τις ερωτήσεις τις έθεσα προς την Κομισιόν, ε, όχι προς εσάς. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι άκουσα το όνομά μου. Ο Ιγνάσιο Γαρσία. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που ετέθεσαν. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση στο Πακιστάν δεν είναι μια απάντηση που βασίζεται αποκλειστικά στο εμπόριο. Αν δείτε στην δήλωση που συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρει ρητά ότι η απάντηση θα πρέπει να ε, συμμορφώνεται και προς την σημαντική ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς και φιλόδοξα εμπορικά μέτρα. Δηλαδή το εμπόριο είναι τμήμα ε, μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης ανταπόκριση σε αυτήν την κρίση που, δια... που περνά το Πακιστάν. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει 320 εκατομμύρια άμεσης ε, ανθρωπιστικής βοήθειας στο Πακιστάν να το αποδεικνύει αυτό. Θα πρέπει δηλαδή αυτό εδώ να το δούμε ως τμήμα μιας ευρύτερης ε, ενό ευρύτερου φάσματο ε, δράσεων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε το Πακιστάν να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεύτερον, ε, αναφέρετε την ανάγκη του Κοινοβουλίου για περισσότερα στοιχεία και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε αυτή η πρόταση πώς ε, επελέγησαν τα προϊόντα, αν έχει γίνει αντίκτυπος οικονομικό και έρευνα για τον αντίκτυπο Φυσικά δεν μπορώ να σας δώσω όλες τις πληροφορίες, αλλά σίγουρα μπορώ να σας δώσω ένα έγγραφο που αναπτύσσει περισσότερο όλα αυτά τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες και όπως είπα ευχαρίστως θα συναντηθούμε με τον εισηγητή για να έχουμε μια πιο λεπτομερή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. η διαφορετική αντιμετώπιση της εθανόλης ε, σε αντιπαράθεση με την κλωστοϊφαντουργία. Η πρώτη μας προσέγγιση ήταν για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα κλωστοϊφαντουργίας. Τα αποκλείσαμε από αυτή την πρόταση, αλλά δεν ε, αποκλείσαμε τη βιοεθανόλη. Καλύπτεται από την πρόταση ακριβώς διότι θεωρήσαμε πως ήταν σημαντικό να συμπεριληφθούν κάποια προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά για την διαφοροποίηση της πακιστανικής οικονομίας. Το θέμα του, την ερώτηση του κυρίου Ζανό την ε, συμβολή που βρίσκεται στη βάση της βιοεθανόλης ε, που εξάγεται από το Πακιστάν. Είναι η μολάσα, η μελάσα, συγγνώμη, είναι δηλαδή ε, παραπροϊόν της παραγωγής ζάχαρης. Δεν σημαίνει δηλαδή την μείωση της διαθέσιμης ζάχαρης προς πώληση στην πακιστανική αγορά. Γιατί το Πακιστάν είναι σημαντικός εξαγωγέας βιοεθανόλης προς την Ένωση και τα επίπεδα που έχουν οριστεί αντιστοιχούν στα επίπεδα εξαγωγών του Πακιστάν κατά το έτος 2008. Και φυσικά όλα όσα θα ε, εξαρθούν υπ' αυτή τη συμφωνία θα ε, είναι υποχρεωτικά σύμμορφα προς ε, την Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το προτιμησιακό κανόνα προέλευσης. Αυτή η προέλευση, αυτός ο κανόνας μπορεί να ανακληθεί και να ανασταλεί η εξαγωγή εάν δεν υπάρχει απόδειξη για την προέλευση αυτής της βιοεθανόλης. Φυσικά και έχω καταγράψει όλε τι παρατηρήσεις του κ. Ζανό και στην περαιτέρω συζήτηση για τα θέματα αυτά ευχαρίστω θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες στα διάφορα διάφορα σημεία που θίξατε. Όσον αφορά τώρα την θέση των τρίτων χωρών στην Γενέβη, εμείς σίγουρα θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες των ΠΟΕ, ώστε να εξασφαλίσουμε υποστήριξη στον ΠΟΕ για την πρόταση αυτή σύντομα. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό είναι ε, ο αντίκτυπος αυτής της πρότασης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε περιλάβει εδώ. Ε, οι συγκεκριμένες αυτές ε, προσανατολισμοί μάλλον μελέτης έχουν εντοπιστεί ως γραμμές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις προτιμήσεις των λιγότερων ανεπτυγμένων ε, των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών και δεν περιλαμβάνονται εδώ. Είμαστε βέβαιοι πως άλλες εξαγωγικές χώρες θα δουν πως υπάρχει ανάγκη να ανταποκριθούμε στο Πακιστάν και από την πλευρά τους να συνεισφέρουν και εκείνες. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν να μπούμε σε παζάρι για το πώς θα αγοράσουμε τη στήριξη άλλων χωρών. Ελπίζουμε πως χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα και άλλες σημαντικές χώρες των ΠΟΕ θα καταλάβουν τη σημασία αυτού του είδους της ανταπόκρισης ιδιαίτερα έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει τώρα το Πακιστάν. Τώρα αναφέρατε διάφορα σημεία που είναι σημεία για θεμητή συζήτηση, διάρκεια, γιατί τρία χρόνια, αλλά κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαφές είναι ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε επενδύσεις, αν θέλουμε να έχουμε βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες για αυτή τη... και μάλλον προς... συγκεκριμένη διάρκεια για αυτή την προτιμωσιακή μεταχείριση, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει αντίκτυπο. Τρία χρόνια ή άλλο ε, διάστημα, δεν ξέρω, μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ, είναι θεμητή συζήτηση αυτή στην Επιτροπή και με τα κρατημέλη, γιατί να σας διευκρινίσω πως πρόκειται για μια πρόταση της Κομισιόν για την ώρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ζήτησε να υποβάλουμε πρόταση, αλλά τα κράτη-μέλη ακόμα την εξετάζουν. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δηλαδή ότι και κάποια κράτη-μέλη θα θέσουν ε, ερωτήσεις για κάποια τμήματα της πρότασής μας. Επίσης ε, λαμβάνω υπόψη τα άλλα θέματα που θίξατε όπως ε, η ρήτρα ε, ασφαλείας, τι θα γίνει με τους δασμούς τους εξαγωγικούς. Το Πακιστάν δεν εφαρμόζει δασμούς για το βαμβάκι και έχουμε υποδείξει στις πακιστανικές αρχές ότι για άλλα προϊόντα μας ανησυχεί το θέμα των δασμών. Είναι πάντως ε, θέματα στα οποία συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πρόταση που θα μπορέσει να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα λεπτομερώς. Να σας πω ειλικρινά πως η Κομισιόν είναι σχετικά σταθερή. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει λόγος να περιορίσουμε τον κατάλογο προϊόντων που έχουμε συμπεριλάβει. Δεν έχουμε πολύ προσεκτικά φτιάξουμε έναν κατάλογο που είναι φιλόδοξος αλλά λαμβάνει και υπόψη τις ευαισθησίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και αν αρχίσουμε να μειώνουμε περισσότερο τα προϊόντα που καλύπτονται από την πρόταση, σύντομα θα φτάσουμε σε μια πρόταση που δεν θα έχει νόημα και δεν θα έχει οικονομικό αντίκτυπο και αξία για το Πακιστάν. Γι' αυτό και κάνω έκκληση να αποφευθεί ο περιορισμός της αξίας των όσων προτείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα. και θα επανέλθουμε σύντομα. Ας προχωρήσουμε στο σημείο... ...8 και 16. Αυτά θα τα εξετάσουμε από κοινού, διότι αφορούν ταυτόσιμες συμφωνίες με διαφορετικές χώρες, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Εγώ είμαι εισηγητής και για τις δύο εκθέσεις αυτές που είναι πολύ παρόμοιες. Απλώς αλλάζει το όνομα της κάθε χώρας. Ζητήθηκε λοιπόν από το Κοινοβούλιο να δώσει τη συνένεσή του στις συμφωνίες ε, που τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες αμοιβέ αναγνώρισης ε, με την ε, Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αυτές οι συμφωνίες αποτέλεσαν την αντικείμενο διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση και απλοποίωση της λειτουργίας της ισχύουσας συμφωνίας η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 1999, δηλαδή πριν 11 χρόνια. Αυτού το είδος οι συμφωνίες είναι συμφωνίες που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης πιστότητας προϊόντων, τα οποία είναι αντικείμενο ρυθμίσεων. Μια τέτοια συμφωνία δίνει σε κάθε ένα από τα συμβαλόμενα μέρη τη δυνατότητα να ελέγχει και να πιστοποιεί προϊόντα σε σχέση με τι κανονιστικέ διατάξει που ισχύουν στο άλλο συμβαλόμενο μέρο, στην επικράτειά του και πριν από την εξαγωγή. Ω εκ τούτου, η Συμφωνία Αμοιβαία Αναγνώριση επιδιώκει να άρει τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, ενώ διασφαλίζει ταυτόχρονα την υγεία, την ασφάλεια και του περιβαλλοντικού στόχου κάθε συμβαλόμενο μέρο. Οι τροπολογίε ε, στο κύριο σώμα της Συμφωνίας ε, έχουν στόχο να επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη δομή των τομεακών παραρτημάτων, να άρουν άσκοπους περιορισμούς ε, εμπορικούς ανάμεσα στους, ε, στα μέρη, να μειώσουν τα διοικητικά βάρη σε σχέση με τη διαχείριση της συμφωνίας και να διευκολύνουν και να διευκρινίσουν τη λειτουργία των συμφωνίων αυτών. Επιπλέον, τα τομεακά παραρτήματα για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές έχουν θεωρηθεί ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις και στις τεχνικές και διοικητικές πρακτικές καθώς και τις αλλαγές που έχουν εισαχθεί από την τροποποιημένη συμφωνία του κύριου μέρους της ε, Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης. Ε, Ενημερώσει για οργανώσει που αναφέρονται και αλλαγές στην νομοθεσία των συμβαλόμενων μερών που επηρεάζουν τον λόγο το με... Ο εισηγητή χαιρετίζει τι βελτιώσει που περιέχονται στις εν λόγω και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινώντα με τη δική μας Επιτροπή, να εγκρίνει τη συμφωνία, τις δύο μάλλον αυτές συμφωνίες. Θα ήθελε κάποιο να πάρει το λόγο για αυτή τη συζήτηση σε συγκεκριτές ήταν αυτή τη φορά ο Κρίστοφερ Φέλντερ και του δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς. Αυτή τη φορά συμφωνείς μαζί μου. Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ και μάλιστα σε βαθμό που νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξετάζουμε τέτοιου είδους εκθέσεις. Γιατί ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται και με πολλά καλά πράγματα, δηλαδή με τους μη δασμολογικούς φραγμούς και ένα, ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει να έρχονται εδώ με εισηγήσει ε, και σκιώδεις εισηγητές. Είναι κάπως τυπικό αυτό το θέμα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να ασχοληθούμε ε, με πολλά σημαντικά αλλά μη επίμαχα ζητήματα και να μην χρειάζεται να κάνουμε μακροσκελή συζητήσει εδώ. Αντί να συζητήσουμε λοιπόν επί της ουσίας, ίσως θα πρέπει εδώ στην Επιτροπή να συζητήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους θέματα στην Επιτροπή μας. Ίσως βέβαια σε κάποιο άλλο φόρμα, αλλά συμφωνώ με τα όσα είπατε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευτυχώ δεν είναι επίμαχα τα θέματα αυτά, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου με την προϋπόθεση ότι θα έρθει εντωμεταξύ σε επαφή μαζί μας το Συμβούλιο. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Άρθουρ Λόπιαν. Μάλιστα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Άρθουρ Λόπιν από την DG Trade. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στην εισηγησή σας. Είπατε όλα τα σημαντικά θέματα, δεν είναι κάτι το νέο. Έχουμε υγιείς σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και απλώς θέλουμε να διευκολύνουμε την διαχείριση και τη ε, διοικητικό ε, σκέλος αυτής της συμφωνίας. Πρόκειται για κάτι τεχνικό, μη ε, αντιφατικό. Ευχαρίστως να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις, αλλά συμφωνώ με τον συγκητή και τον σκιώδη συγκητή. Σας ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτών των θεμάτων. Το επόμενο θέμα είναι δηλαδή απόψεων με τον αρμόδιο για το εμπόριο επίτροπο Κάρελ Ντε Κούχτ που έχει προγραμματιστεί για τις 5 και ε, από ό,τι φαίνεται θα φτάσει στην ώρα του στις 5. Δηλαδή κάπως προχωρήσαμε πολύ γρήγορα, ε, ασυνήθιστα γρήγορα προχωρήσαμε. Γι' αυτό και θα διακόψουμε μέχρι τις 5. Σας ευχαριστώ όλους. Ελάτε φίλε και φίλοι, ας συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας. Καλωσορίζω και πάλι τον Επίτροπο Εμπορίου Κάρελ Ντεγκούχτ. έχουμε ορισμένα θέματα σημαντικά στην ημερήσια διαταξή μας. Το μέλλον της εμπορικής πολιτικής, της προτιμήσεις υπέρ του Πακιστάν, αν και τα έχουμε συζητήσει αυτά πιο πριν, τις διαπραγματεύσεις άκτα, την πολιτική αλλοδαπών επενδύσεων της Ένωσης και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο. αρχίζει και γίνεται πια τακτικός επισκέπτης στις συναντήσεις μας ο κύριος Επίτροπος. Και θα προχωρήσουμε σε καρποφόρο ανταλλαγή απόψεων με τον ίδιο. Εάν έχουμε αρκετό χρόνο και αν θεωρεί και ο ίδιος ότι είναι σκόπιμο, θα ήθελα να προσθέσουμε και τις της Μερκοσούρ Βέβαια θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο. Μετά από τον Επίτροπο θα λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επίτροπε που ήρθατε και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ζητώ πρώτα συγγνώμη για την καθυστέρηση της αφήξεώς μου. Η επίσκεψη του Γενικού Διευθυντού του ΠΟΕ του κ. Πασκάλ Λαμί. έγινε και αυτή με κάποια καθυστέρηση έτσι λοιπόν η μία καθυστέρηση έφερε την άλλη ανάμεσα στις δύο αυτές ανειδημένες υποχρώσεις μου στο Στρασβούργο διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλειά σας συζητήσεις για τα τρία θέματα την προηγούμενη Τετάρτη, ίσως και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωβουλής, μια ολόκληρη βραδινή συνεδρίαση είχε αφιερωθεί σε θέματα εμπορίου, αν και όλοι θα προτιμούσαμε βέβαια να είμαστε σε ένα συμπαθητικό εστιατόριο στην πόλη αυτή. Η εμπορική πολιτική πάντως έχει σημασία και αυτό το αντιλαμβάνεται βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να επανέλθω διαμακρών στα θέματα που συζητήθηκαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, για το Πακιστάν και τη συμφωνία Άκτα θα πω ωστόσο λίγα λόγια εφόσον πρόκειται να τα συζητήσετε αυτά τα θέματα και τις προσεχείς εβδομάδες. Χαίρομαι για την πρόθεση που έχετε να προχωρήσετε ταχαίως σε συζητήσεις για τα θέματα αυτά για να έχουμε την ε, βάση για μια ε, βιώσιμη ανάπτυξη του Πακιστάν. Ήδη συζητήσατε με την Γενική Διεύθυνση ε, ε, Εμπορίου τη δική μας για το Πακιστάν. Ευχαριστώ να απαντήσω σε ε, ερωτήσεις που ίσως έχετε ακόμη. Σε ό,τι αφορά την συμφωνία Άκτα, επαναλαμβάνω τα όσα είπα την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος της συζητήσεως, ότι δηλαδή χρειάζεται μια συζήτηση βασισμένη σε πληροφόρηση. Και βεβαίως είστε ε, ευπρόσδεκτοι να μου υποβάλλετε οποιασδήποτε παρατηρήσεις ή σχόλια έχετε σχετικά με την συμφωνία. Να δούμε και πού ακριβώς διαφωνούμε. Δηλαδή, ε, στην ε, ανάπτυξη της... Μάλλον που συμφωνούμε στην διαμενάδηση της Ένωσης βασισμένη σε μια κοινωνία της γνώσης. πράγματα που θα περιλάβουμε και στην ανακοίνωσή μας για την Ευρώπη 2020 που θα υποβληθεί αρχάς Νοεμβρίου. Χαίρομαι για την απόφαση της Επιτροπής σας να αναλάβει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και για την συζήτηση που θα γίνει μετά από την ε, διαβίβαση αυτής της εκθέσεως. Ό,τι αφορά το μελλοντικό μας έργο, δύο θέματα θα μας απασχολήσουν. Πρώτον, οι μελλοντικέ ε, ρυθμίσεις του Γενικού Συστήματος Προτιμήσεων, του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διεξάγει τώρα μελέτη επιπτώσεων, μελέτη αντικτύπου. Μετά από την έγκρισή της ΔΕ σε λίγες εβδομάδες η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Ευρωβουλή. Στις αρχές του 2011 η Κομισιόν θα σας υποβάλει έκθεση για την πρόοδο των κυρώσεων της συμφωνίας αυτή επίσης κατάλογο των χωρών που εποφελούνται, καθώς και τις σχετικές ε, συστάσεις των αρμόδιων οργάνων. Θα είμαστε πλέον σε θέση να υποβάλουμε πρόταση για ένα μηχανισμό διαδοχής. Το πρώτο ήδη τρίμηνο, ήδη τρίμηνο του 2011 ώστε το σύστημα ε, γενικευμένων προτιμήσεων να γίνει πιο απλό και κατανοητό. με ιδιαίτερη στόχευση πρώτο να, να ε, πάνε τα ωφέλη κυρίως σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από τις χώρες αυτές δηλαδή να γίνει μεγαλύτερη, ε, να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση του μηχανισμού που να επιτρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέρη στις ε, προτιμήσεις αυτές. Τρίτο, το νέο θεσμικό πλαίσιο με μεγαλύτερη εμπλοκή επομένως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, εγώ σημείωσα τις ανησυχίες της Επιτροπής σας που διατύπωσε στην επιστολή του ο Πρόεδρός σας τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε δηλαδή. Και αναμένω την απάντηση στην ανακοίνωση πολιτικής μας που κάναμε τον Ιούλιο σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να λησμονούμε και το χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διαπραγματεύσεις με Καναδά, Ινδία και Σιγκαπούρη για την προστασία των επενδύσεων που είναι θέμα πρώτης της σημασίας και προς το συμφέρον βέβαια των συνολικών μας εμπορικών σχέσεων. Πρέπει επομένως να διατηρήσουμε την ε, ε, πρόοδο της, ε, των διαπραγματεύσεων αυτών και για τις σχέσεις βέβαια μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Θα στείλουμε τις τελευταίες τροποποίησεις των διαπραγματευτικών οδηγιών με τις χώρες αυτές. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, οι διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις Τροποποιητικέ αυτέ οδηγίες θα γίνουν μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που να μας επιτρέψει να αρχίσουμε ουσιώδεις συζητήσεις με τους εταίρου μας ήδη από τις αρχές του επόμενου χρόνου, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελλοντική πολιτική επενδύσεων με τις τρεις αυτές χώρες. Ένα άλλο θεσμικό θέμα είναι η επιτροπολογία. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές, να μην υπάρχει δηλαδή αμφιβολία σχετικά με τις απόψει μου. Η επιτροπολογία θα πρέπει να υπακούει στους συνήθεις κανόνες επιτροπολογίας χωρίς μεταβατικές περιόδους. Βρισκόμαστε στον χώρο της τακτικής, της συνήθους δηλαδή νομοθετική διαδικασίας, χωρίς εξαιρέσεις. Η Κομισιόν θα το εξασφαλίσει αυτό αφενός στον κανονισμό στον οριζόντιο κανονισμό επιτροπολογία, καθώς επίσης και σε ειδικέ πράξει τις οποίες θα σα υποβάλουμε σύντομα και αναμένω την υποστήριξή σας. Θα ήθελα με την ευκαιρία επίσης να ανακοινώσω ότι θα γίνει συζήτηση ή μάλλον ε, η ημερομηνία θα είναι 17 Δεκεμβρίου για την επόμενη συνάντηση ΤΕΚ. Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να βρούμε ημερομηνία πριν από την διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκής Ένωση Ενωμένων Πολιτειών. Αλλά θα είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους ηγέτε μας για να μπορέσουν να διαπραγματευτούν τα ΤΕΚ που είναι ε, σημαντικό, σημαντική βάση για τη συνεργασία και χρειάζεται περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα από ό,τι στο παρελθόν. Για την καλύτερη ολοκλήρωση της διατλαντικής αγοράς. για να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις της καινοτομίας και μιας πιο, μιας πιο πράσινης οικονομίας και οι προκλήσεις σημαντικών νέων αναπτυσσόμενων οικονομιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εν μια νυχτή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε απέναντι στις ΗΠΑ και εν τέλει το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχετε αύριο στην ημερήσια διαταξή σα, έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να κινηθεί μέσα σε ένα κενό. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κοινωνιών. Η πρόκληση για μα είναι να επιτύχουμε να λειτουργεί το εμπόριο λαμβάνοντας υπόψη τις θεμητές αυτές ανησυχίες. Το εμπόριο πάντως ήδη έχει παίξει σημαντικό, αλλά, σημαντικό ρόλο που δεν έχει όμως αναγνωριστεί πλήρως για την αύξηση των βιωτικών επιπέδων. Η εμπορική πολιτική έχει δώσει επίσης σημαντικά κίνητρα και αντικίνητρα βεβαίως για την συμμόρφωση με τις διεθνείς ε, συμφωνίες. Ας παραμείνουμε ρεαλιστές σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ε, να υπάρξουν άλλα επιτεύγματα. Ας μην βάλουμε πολύ ψηλά τους στόχους για να μην απογοητευτούμε. Η εμπορική πολιτική δεν είναι ένα οποιοδήποτε εργαλείο. Επίσης η εμπορική πολιτική υποτίθεται ότι εξυπηρετεί και άλλους στόχους και βεβαίως και την ευημερία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και, και εγώ κύριε Επίτροπε. Ας ακούσουμε τώρα τους προσώπους των πολιτικών ομάδων και θα αρχίσουμε με το Λαϊκό Κόμμα. Βλέπω ότι ορισμένα, ε, διάφορα μέλη μάλλον της Επιτροπής θέλουν να λάβουν το λόγο, άρα θα επιβάλλω χρονικό όριο το, στις αγορεύσεις. Ε, εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Κουίστχαουτ Ρόβολ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Με συγχωρείτε. Θέλετε να μιλήσω γαλλικά, αυτό είναι. Α, όχι, όχι, απλώς ζητώ το λόγο, κυρία μου. Και γαλλικά μπορώ να μιλήσω, συνεχίζει η κυρία Ρόβερ. Έχει καλώ. Συνεχίζω στα γερμανικά. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον Επίτροπο που προσέρχεται τακτικά στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας με, σε, με σάρκα και οστά. Μια πρώτη ερώτηση εξ ονόματος της ομάδος μου. Τονίζεται ότι θα ε, μεταχειριστείτε την επιτροπολογία και στο εμπόριο με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που και στους άλλους τομείς. Εσείς ε, λέτε ότι αυτό είναι απόλυτα σίγουρο, μα το εμπόριο δεν είναι ένας τομέας όπως η συνήθις τομή των της εξωτερικής πολιτικής, των εξωτερικών σχέσεων. Βρίσκεται σε ένα είδος interface ανάμεσα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Κάπου βρίσκεται λοιπόν ενδιάμεσα. Εγώ ε, και εγώ το βλέπω έτσι, αλλά και η πολιτική μου ομάδα βλέπει ότι υπάρχουν διαφορές. Νομίζω ότι μπορεί ωστόσο ή πρέπει να αναζητηθεί μια ρεαλιστική δυνατότητα ε, συνεργασίας. Επίσης, αναφερθήκατε σε διάφορες διμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύεστε ήδη διμερός. Δεν έχω ακούσει όμως από εσά τελευταία τίποτε σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν άκουσα καλά όμως πριν μιλήσατε ήδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΠΟΕ, κύριο Λαμί. Βλέπετε τώρα την δυνατότητα όταν λήξει ο γύρος της Δόχα, μάλλον βλέπετε να λύγει κάποτε ο γύρος της Δόχα, εδώ και χρόνια μας απασχολεί. Και δεν είμαι βεβαία ότι πράγματι είναι ο καλύτερος ε, δρόμος προς το μέλλον. Τέλος, σε μια μάλλον ας πούμε ανεπίσημη συζήτηση με Αμερικανούς τονίστηκε πάλι για πολλωστή φορά ότι οι Ενωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη συμμερίζονται μεν τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες και θα έπρεπε να διαπραγματεύονται από κοινού διάφορες ε, συμφωνίες. Πώς βλέπετε τις δυνατότητες αυτές, για παράδειγμα απέναντι στην Κορέα, απέναντι σε άλλες χώρες. Πώς βλέπετε τη δυνατότητα δηλαδή να διαπραγματευτούμε στο πλευρό των Αμερικανών. Δεν θα ενίσχυε κάτι τέτοιο την θέση της Δύσεως συνολικά. Τώρα ο κύριος Καντέρα Ρίφ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για ένα σημείο το οποίο ανέφερε το θέμα της Επιτροπολογίας, όχι τόσο γι' αυτό, αλλά τον ευχαριστώ γιατί ε, ξέφρασε έντονα τη θέση του για την ε, θέση του Κοινοβουλίου και με ευαισθητοποιεί το γεγονός ότι υποστηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου η Κομισιόν. Κυρίως όταν βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία διάθεση να προχωρήσουν και τείνουν να παριστάνουν πως η συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχει και ότι το θέμα της εμπορικής πολιτικής είναι δικός τους, ε, δική τους υπόθεση αποκλειστικά. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ ε, και μπορείτε να βασιστείτε σε εμά, εκφράζομαι στο όνομα της ομάδας μου, ε, ότι θα σας στηρίξουμε σε αυτήν ε, την υπόθεση. Για να μιλήσω γρήγορα, για το Πακιστάν δεν είχα την ευκαιρία και ζητώ συγγνώμη να συμμετέχω στη συζήτηση που έγινε πριν από λίγο. Κάποιες, κάποιοι προβληματισμοί. Μια χώρα που ήδη εξάγει 900 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κλωστοϊφαντουργία. Προσθέτουμε και 5 επιπλέον εκατομμύρια με ένα μεγάλο, μεγάλο φόβο ε, στις ευρωπαϊκές αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι αυτό έχει αντίκτυπο και σε τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις, όπως ε, οι χώρες της Νοτίου όχθης της, Αμερι... της Μεσογείου ή με την Τουρκία. Είχαμε κάνει μια συνεδρίαση αντίστοιχη όταν ανοίξαμε την αγορά μας στην ε, Κινέζικη κλωστοφαντουργία πριν από λίγα χρόνια. Γιατί λοιπόν αυτός ο κανονισμός για τρία χρόνια θα μπορούσε να ισχύσει για ένα ή δύο χρόνια. Δείτε, ε, η κατάσταση είναι υπό εξέλιξη. Τρία χρόνια είναι μια συμφωνία γενικευμένων προτιμήσεων συν για το Πακιστάν καμουφλαρισμένη. Ενώ σε τρία χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε ε, διαβλέψει, προβλέψει μια τροποποίηση του κανονισμού για να δούμε αν τελικά το Πακιστάν θα μπορούσε να ε, ωφεληθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα, στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο εκφράσαμε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Λέτε ότι δεν αλλάζει τίποτα για αυτό το θέμα για την ώρα. Υπάρχουν όμως κάποιοι προβληματισμοί για το γεγονός ότι διατηρούμε το θέμα των όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε <laughs> λες και παίζουμε το παιχνίδι των, ε, της μουσικής ε, καρέκλας. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος σταματά και δεν είναι ένα ε, ρυθμισμένο δικαίωμα, γιατί μπορεί να τιμωρηθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει να εμπορευτεί. Τώρα, νομίζω σας είχα θέσει το ερώτημα αυτό. Σε τι χρησιμεύει κάτι τέτοιο και γιατί το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ο βασικός προβληματισμός. Δεν υπάρχει καμιά πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Για τις επενδύσεις είναι πράγματι ένα νέο θέμα για μας, ένα πακέτο επενδύσεων που αφορά από τη μια πλευρά τον κανονισμό και από την άλλη μια ανακοίνωση. Εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι συγγετής για το θέμα αυτό και είμαστε μόνο στην αρχή. Αλλά βεβαίω ακούμε όλα τα ερωτήματα που τίθενται τη σήμερα ημέρα, δηλαδή το θέμα τη αμοιβαιότητα. Ποια είναι η δική σα επεπίθεση και η ανάλυση σα για το θέμα αυτό. Τώρα, το θέμα ανάλογα με τη χώρα. Είναι μια συζήτηση αυτή στα κρατημέλη. Το θέμα, α πούμε, των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι η απόφαση του ΔΕΚ που, στην οποία βασιζόμαστε ή είναι κάποια άλλη ερμηνεία ας πούμε, τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων που έχει επιπτώσεις στα κράτη, μεγάλες μάλιστα. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Επίσης, αν είναι μόνο οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν δικαίωμα να στραφούν στο όργανο διευθέτησης διαφορών, μήπως θα μπορούσαν και τα κράτη, τα συνδικάτα να στραφούν προς εκεί. Έχω πολλά ερωτήματα, αλλά ήθελα απλώς να σας δώσω μια ιδέα για το ποιους προβληματισμούς έχουμε, κύριε Επίτροπε, για το θέμα των επενδύσεων, για τις ε, διατλαντικές σχέσεις. Βλέπω το σημερινό κείμενο, σήμερα το ανακαλύπτουμε. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν κάποια θετικά ε, μηνύματα θα ήθελα να ξαναμπεί ο, η ρύθμιση διαφορών, ας πούμε όπως αυτή η υπόθεση της Boeing, το θέμα της δημόσιας υγείας όταν λέμε για αμοιβαίο σεβασμό, κάτι τέτοιο αφορά τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τις ορμόνες και ένα σωρό άλλα ε, θέματα και ποια είναι η θέση των Αμερικανών επ' αυτών. Και τέλος, για την ανακοίνωση για τη νέα εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το λέω εγώ, αλλά πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν ήταν επιτυχής και να μπω στην σε κάποιες λεπτομέρειες. Ε, το βλέπω και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί το υπερασπίζομαι το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής μέσα στους προβληματισμούς της Κομισιόν. Ναι, ναι, ολοκληρώνω και ταυτόχρονα υπογράφουμε ένα σωρό συμφωνίες. Ε, έχουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη υπογράφει όλες τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών από τη στιγμή που κάποια χώρα τη το ζητά, χωρίς να προβληματίζεται. Ας πούμε για την Νότιο Κορέα που αφορά τις υπηρεσίες δεν μετρούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, ας πούμε, για την απασχόληση. Αυτά σύντομα. Αυτή σύντομα ήταν η προβληματισμή μου. Ε, ε, έχουμε τώρα μόνο μια ώρα στη διάθεσή μας. Παρακαλώ λοιπόν, σας ζητώ από τους ομιλητές να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. δεν είναι ερωτήσει. αυτό είναι μια, ένας κατάλογος των όσων μπορούν να συμβούν στο εμπόριο. Γιάννη Ζανό, των Περσίνων. Με συγχωρείτε. Έχουμε καταρχήν τους φιλελεύθερους οι οποίοι έχουν ε, ζητήσει το λόγο, Μαρία Σαρνές. Μην ανησυχείτε. Δεν θα μιλήσω περισσότερο χρόνο από ό,τι προλαλή σα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό, σα το υπόσχομαι. Εγώ θα ήθελα απλώ να θέσω κάποιε ερωτήσει πολύ συγκεκριμένε για το ΑΚΤΑ, για τη συμφωνία λοιπόν αυτή που θα υπογράψουμε. Νομίζω ότι εδώ ε, υπάρχει κάτι που βλάπτει το περιεχόμενό του και αυτό είναι το θέμα του απορρίτου. Γιατί αυτή τη στιγμή ακούγονται πάρα πολλές φήμες γύρω-γύρω και αυτό που προσπαθούμε εμείς είναι να επιβάλλουμε τη διαφάνεια. Αυτό χρειάζεται. Γιατί βέβαια υπάρχουν τα θέματα των ατομικών δικαιωμάτων, το διαδίκτυο, όλα αυτά κινητοποιούν και πολύ σωστά την κοινωνία, αλλά βέβαια τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα προβλήματα της ε, παραποίησης κτλ. Είναι θέματα τα οποία ξεπερνάνε το διαδίκτυο. Ε, αυτή πρόσφατα είχα πάει στην ε, Νότιο Κορέα και ξέρετε τι έγινε ε, με τη Samsung και το iPad. Έχει απαγορευτεί κάθε εισαγωγή του iPad στην Νότιο Κορέα μέχρι η Samsung να φτιάξει το δικό της μοντέλο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά λοιπόν τα, το μυστήριο, τα ενίγματα, το απόρριτο είναι θέματα τα οποία καλό θα τα να αφήσουμε στην άκρη. Τώρα, σχέση με Μερκοσούρ, συμφωνία. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό, το οποίο ψήφισε την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο στο γνωστό ψήφισμα για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων όπου οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, της ανθρώπινης υγείας κτλ. πρέπει να γίνονται σεβαστές. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε νομολογία αντίστοιχη, η οποία μετά θα ισχύει για κάθε συμφωνία εμπορική πολιτικής. Εγώ νομίζω ότι η αμοιβαιότητα για την οποία συζητάμε τόσο πολύ ε, θα έπρεπε να λαμβάνει αυτέ τι πτυχέ υπόψη. Πείτε μου εσεί λοιπόν αυτή τη θέση του Κοινοβουλίου πώ θα τη λάβετε υπόψη στι μελλοντικέ σα διαπραγματεύσει για το Μερκοσούρ. Τρίτον, Πακιστάν. Βεβαίω το θέμα της κλωστοϊφαντουργίας ε, και της εθανόλης που θα θίξει ο συνάδελφος τώρα που θα πάρει το λόγο. Ξέρω ότι όλα αυτά ανησυχούν τους Ευρωπαίους. Όμως αναγνωρίζω την αναγκαιότητα μιας μάλλον πρωτότυπης συμφωνίας με το Πακιστάν. Γιατί χρειάζεται να έχει πολύ θετική ε, θετικές επιπτώσεις για τους ίδιους τους Πακιστανούς, για το λαό. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση έτσι ώστε για την ευημερία των κατοίκων αυτής της περιοχής η συμφωνία αυτή να φέρει θετικά αποτελέσματα. Και τελευταίο και τέταρτο, όσα είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, οι εμπορικές σχέσεις. Πώς θα εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητας, την οποία τόσο συζητάμε, μια και δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται πουθενά στην πράξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντό, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αφού μου ζήτησε συνάδελφος να πω δύο λόγια για την εθανόλια, ε, θα τα πω. Λοιπόν, κατανοείτε ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερα το κεφάλαιο αυτό. Στο σχέδιο έκτακτης ε, βοήθειας που προτείνεται για το Πακιστάν και εκπλήσωμαι που σε ένα σχέδιο το οποίο έχει ως στόχο να, στηράξει, να στηρίξει με συγχωρείτε, τους Πακιστανούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλά θέματα διατροφικής ανασφάλειας, ασχολούμαστε με ένα βιοκαύσιμο. Και τα βιοκαύσιμα, ξέρετε, καλλιεργούνται πάντα στη θέση άλλων παραδοσιακών καλλιεργιών τροφίμων. Είμαι κάπως εκνευρισμένος, γιατί εγώ φανταζόμουν πως θα έρθετε εδώ να μας παρουσιάσετε λίγο τα έγγραφα της 9 η Νοεμβρίου, τη στρατηγική, την εμπορική ε, στα πλαίσια της Ευρώπης του, 20, του 2020 και είδα ότι ήσασταν πολύ ολιγόλογος στο θέμα αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε κάτι παραπάνω, να μας πείτε και ποιος είναι ο απολογισμός που θα κάνετε του Global Europe. Γιατί και οι προηγούμενοι συνάδελφοι το αξιολόγησαν μάλλον αρνητικά. Ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα για τη νέα στρατηγική που θα χαράξετε και πώς έχετε σκοπό σε μια συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων που είναι αρκετά σκληρή σήμερα πολλές φορές για τα εξαγωγικά μοντέλα. Πώς θα εντάξετε λοιπόν την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Γιατί βέβαια αυτή στηρίζεται σε κάποιες εσωτερικές ισορροπίες. Έχουμε το εξωτερικό μοντέλο της Γερμανίας, το οποίο πολλές φορές αμφισβητείται από την Ευρώπη σήμερα. Να δούμε λοιπόν τι προοπτικές βλέπετε εσείς. Θα δούμε τι θα πει και G20 στο Pittsburgh για να ισορροπήσουν λίγο οι σχέσεις Κίνας-Ευρώπης, είπα. Να δούμε λοιπόν αυτό τι θα σημαίνει για την εσωτερική δυναμική που κινεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για τη δομή που θα δώσουμε στι εξαγωγικέ μα προσπάθειε. Να μην είναι λοιπόν πάντα ε, ασαφή αυτά και τις κλιματικές ε, τα κλιματικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πώς θα τα εντάξετε και αυτά στις εμπορικές πολιτικές του μέλλοντος. Σόλτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Πίτροπε. Ήδη με έχουν καλύψει ορισμένοι συνάδελφοί μου με τις ερωτήσεις που έθεσαν. Έχω λοιπόν ακόμα τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μιλήσατε πρώτα, είπατε για την ε, ημερομηνία της επόμενης συνάντησης των ΤΕΚ. Ποιες όμως θέσεις θέλετε να υποβάλλετε σε αυτήν την συνάντηση και ποιο είναι το νόημα αυτής της νέα συνάντησης των ΤΕΚ για τις προκλήσεις, παγκόσμιες προκλήσεις και πώς βλέπετε τις διμερείς σχέσεις με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και πώς αυτές οι σχέσεις διαμορφώνονται μέσα σε ένα πολυμερές περιβάλλον. Δεύτερο, η αίτηση του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου ε, στη συνάντηση αυτή ΤΕΚ. ώστε να προκύψει και μεγαλύτερη διαφάνεια και υπέρ του Κοινοβουλίου και υπέρ του Κόγκρεσου. Επίσης, άκουσα τα όσα είπατε για τη Συμφωνία Άκτα στο Στρασβούργο. Διάβασα όμως και τα ψηλά γράμματα. που εμείς οι Γερμανοί πάντα τα προσέχουμε τα ψηλά γράμματα. Και υπάρχει μια υποσημείωση υπαριθμών 2 για ένα από τα ανοιχτά θέματα που λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να αποκλείσουν τις ευρεσιτεχνίες από την συμφωνία. Αυτό συνδέεται με την συζήτηση και αποναφέρεται και στα χωρίς ε, εμπορική ονομασία φάρμακα. Εδώ ανοίγεται ένας δρόμος για να εισχωρήσουν αντιφάσεις στη συμφωνία. Τέλος, πάλι για την Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορικών Ανταλλαγών μεταξύ Ένωσης και Ινδίας για τα δεδομένα κλινικών δοκιμών να περιληφθούν δηλαδή στην συμφωνία γιατί οι εταιρείε οι οποίες παράγουν ε, φάρμακα του generic, δηλαδή χωρίς εμπορική ονομασία, ε, είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή, δέχεστε να βγάλουμε την αποκλειστικότητα των δεδομένων από το κείμενο της ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών μεταξύ Ένωσης και Ινδίας. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Επανέρχομαι στα όσα είπε ο πρώτος ομιλητής σχετικά με το ανοιχτό πνεύμα και τη διαφάνειά σας. Κάποιος είπε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέρευσε λόγω των κακών της τρόπων. Δεν θα μπορούσε ποτέ να πει κανείς κάτι τέτοιο για σας. Βέβαια κύριε Επιτροπέ. Θα είμαι σύντομος. Μία από τις συνέπειες της συνθήκης Λισαβόνας είναι η συμμετοχή σε συναπόφαση του Κοινοβουλίου και για εμπορικές συμφωνίες. Η διαφάνεια λοιπόν είναι καταρχήν καλό πράγμα και οι επιπτώσεις της είναι πάντοτε θετικές. Όσο περισσότερη διαφάνεια ε, υπάρχει, τόσο πιο καλές και στέρες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος και μάλιστα σημαντικός και βλέπουμε πολλά παραδείγματα και στην Επιτροπή μας εδώ. Το τα λέω εγώ στους συναδέλφους μου. Την πολιτικοποίηση δηλαδή της εμπορικής συμφωνίας που δεν είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή να υπάρξει τέτοια πολιτικοποίηση της εμπορικής πολιτικής. Εμείς θέλουμε και ο Ευρωπαίος καταναλωτής θέλει να υπάρχει ακεραιότητα στην ε, εμπορική πολιτική και ίσως εσείς κύριε Επίτροπε, θα μπορείτε να είστε ο θεματοφύλακα τη ακαιρεότητα αυτή στην εμπορική πολιτική. Τώρα, δύο πολύ σύντομα σχόλια για τι χώρε τη κοινοπολιτεία. Δύο από αυτέ που είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Βρετανία, αλλά και για το κόμμα μου. Για τις προτάσεις ε, υπέρ του Πακιστάν, εμείς είμαστε υπέρ και με την ευκαιρία αυτή θα πω στους ε, συναδέλφους μου εδώ της Επιτροπής θα τους ε, συστήσω να υποστηρίξουν. Θα πω στον κύριο Αρίφ, νομίζω ότι ήταν ο κύριος Αρίφ ότι ο λόγος που επιλέχθηκε η τριετία είναι ότι ένας χρόνος προτιμήσεων δεν ε, ισοδυναμεί σχεδόν με τίποτα. Τρία χρόνια είναι 8-9 φορές περισσότερος όγκος ε, των συναλλαγών από ένα χρόνο. Πολύ ευχαρίστως να συζητήσω πάντως τα πράγματα αυτά με τους συναδέλφους μου και να εξεύρουμε και χώρο συνεργασίας και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα να πω κάτι και για την σκληρή μεταχείριση κάτι τη Σρι αλλά θα το αφήσω για την ώρα αυτή. Ένα τελευταίο σχόλιο, κρίμα που δεν είναι ο Τζοε Higgins εδώ, θα πω δηλαδή ότι αναπτύσσεται κριτική από την αριστερή πλευρά, η οποία λέει ότι οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν εν τέλει σε ένα κρυφό dumping των αγροτικών προϊόντων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, βλάπτοντας έτσι τους ε, παραγωγούς των ε, αναψώμενων χωρών. Αυτό το έχει πει εύγλωτα ο Higgins σε προηγούμενη ε, συνεδρίαση. Και ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν έκανε σαν να μην είχε ακούσει ποτέ. Ενώ μια κριτική που ασκείται εδώ και τρει δεκαετίε. Εμεί έχουμε σημαντικέ ανησυχίε για το θέμα αυτό. Θα παρακαλέσω τον Επίτροπο, παρόλε τι πολλέ υποχρεώσει που έχει σε άλλου τομεί, να εξετάσει προσεκτικά τον τομέα αυτών των επιδοτήσεων υπέρ των αγροτικών προϊόντων της Ένωσης και τις επιπτώσεις που έχουν οι εξαγωγές αυτές στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μάλιστα, εδώ λίγο ο πρώτος γύρος, κύριε Επίτροπε. Ε, έχουμε ήδη φτάσει 6 παρα 10 και έχω ακόμα 3 εγγεγραμμένους. Νομίζετε ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο και στους εναπομένοντες. Μου, μου έχετε ήδη υποβάλει καμιά 25 ερωτήσεις από ό,τι βλέπω. Να, μόνο αυτές που υπέβαλε ο κύριος Αρίφ είναι σαν το λαρούς, το λεξικό. Ας αρχίσω και θα δούμε. Επιτροπολογία, κυρία Κουίσταουτ. Ίσως να αληθεύει εν μέρη ότι το εμπόριο εμπεριέχει πολιτικά στοιχεία. Από τη μια πλευρά είναι γεωστρατηγική σημασία, ιδιαίτερα με κάποιους εταίρους. Από την άλλη πλευρά είναι ένα πολυτεχνικό ζήτημα. Και βέβαια η οικονομική του σημασία είναι ξεκάθαρη θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μακροσκελή συζήτηση από αυτό. Πάντως το θέμα είναι ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι σαφές ότι δεν γίνεται διάκριση για το εμπόριο. Είναι απλό το πράγμα. Καθώς διτέλεσα δικηγόρος ε, για 25 χρόνια, πάντοτε μπορώ, ε, μπορώ να βρω ένα επιχείρημα. Πάντως η συνθήκη είναι αυτή που συμφώνησαν τα κράτη-μέλη και η Γερμανία και είναι ξεκάθαρο εκεί. Δεν γίνεται καμιά διάκριση για το εμπόριο. Πέρα από αυτό συμφωνώ ότι εμπεριέχει ένα πολιτικό στοιχείο και αυτό είναι και που με ευχαριστεί κιόλας στο εμπόριο. Ο ΠΟΕ. Μόλις ε, είχα μια συζήτηση με τον Πασκάλ Λαμή, τον βλέπω αρκετά συχνά και του μιλάω συχνά και στο τηλέφωνο. κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση για την Τόχα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε τους Αμερικανούς μας εταίρους ώστε να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν είναι εύκολο να ξέρει κανείς τι έχουν στο μυαλό τους. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο μέχρι να μας πούν όταν θα έχουν περάσει οι εκλογές και θα είναι ξεκάθαρη η πολιτική τους επιλογή. Πάντως συμφώνησαν ότι θα ξανασυζητηθεί το θέμα στη Σεούλ στη G20. Παλιότερα ήταν πολύ διστακτική, ενώ τώρα όχι. Και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ξεκάθαρη ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα πρόταση να διαπραγματευτούμε από κοινού με τους Αμερικανούς. Εγώ το έχω ήδη προτείνει ότι θα μπορούσαμε για παράδειγμα να το κάνουμε αυτό σε σχέση με μια συμφωνία επενδυτική με την Κίνα. Δεν είναι νομίζω δυνατόν για συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών γιατί προφανώς εκεί μπαίνει το θέμα του ανταγωνισμού. Και τουλάχιστον μέχρι τώρα είμαστε σε θέση στην Ευρώπη να παρουσιάζουμε τις συνθήκες τις οποίες έχουμε διαπραγματευτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη ΣΥΠΑ, αν και έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Νότιο Κορέα, την Κολομβία και τον Παναμά πριν από λίγα χρόνια, δεν τις έχουν ακόμα παρουσιάσει. Νομίζω όμως ότι για μερικά θέματα είναι λογικό. Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με πιθανή επενδυτική συμφωνία με την Κίνα θα είχε νόημα, αλλά βέβαια αυτό θα αποφασιστεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Τώρα, οι ερωτήσεις ε, του Καντέρ Αρίφ. Θα είμαι γνώμων που συμφωνείτε μαζί μου με την, για την επιτροπολογία, κύριε Αρίφ, αλλά έχω την εντύπωση ότι διαφωνείτε σε όλα τα άλλα. Αλλά, μπας περιπτώσει, κάτι είναι και αυτό. Γιατί τρία χρόνια για το Πακιστάν. Γιατί θα πρέπει αυτό αυτή η συμφωνία να ενταχθεί σε έναν εμπορικό κύκλο. Και εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε για την τύχη του Πακιστάν στο επόμενο πρόγραμμα γενικών προτιμήσεων. Δηλαδή είναι στα χέρια σας. Έχετε στόχο να το συμπεριλάβετε ή όχι. Εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε για την άκτα. Εδώ πραγματικά πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Είμαι επίτροπος για το εμπόριο εδώ και 8 μήνες και έχουμε κάνει τρεις συζητήσεις στην Ολομέλεια για το ΆΚΤΑ. Πάντα τις ίδιες ερωτήσεις μου κάνετε και δίνω τις ίδιες απαντήσεις πάντα. Που δεν επιδέχονται επικρίσεων γιατί είναι πράγματα προφανή. όλα αυτά διαρκώ τι ίδιε ερωτήσεις μου υποβάλλετε. Και ακόμα μια φορά σήμερα εσείς και η κυρία Ντεσσαρνέ για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Εδώ έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά, γιατί υπήρχε σαφής άρνηση των Αμερικανών όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ενώ τώρα η αρχή της νομιμότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων έχει εγγραφεί και το ίδιο για το border enforcement. Ε, υπάρχει η συμφωνία επί της αρχής. Πολύ μεγάλο βήμα μπροστά έχουμε κάνει. Αν πιστεύετε πραγματικά πως είναι δυνατόν να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς απόλυτη ισότητα για τις γεωγραφικές ενδείξεις, προτείνω να σας ορίσω απεσταλμένο μου για να το διαπραγματευτείτε εσείς μαζί τους. Πραγματικά Έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να πιέσουμε τους Αμερικανούς για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Και νομίζω πως το αποτέλεσμα δεν είναι κακό. Τώρα, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε ευρεσιτεχνίε και τα φάρμακα χωρίς εμπορική ονομασία. Η άκτα είναι σαφής για το, αυτού του είδου τα φάρμακα. Διμερή συμφωνία μας ε, με την Ινδία θα είναι επίση ξεκάθαρη. Γίνεται αυτή τη στιγμή συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ινδίας και Βραζιλίας για το τι θα πρέπει να γίνει. Νομίζω πως ε, προχωρούμε προς μια συμφωνία. Είναι αλήθεια πως υπήρξαν προβλήματα, κυρίως για μια χώρα μέλος που σταμάτησε τις μεταφορές που ήταν σε τράνζιτ. Αλλά δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος από αυτό. Εγώ νομίζω πως είναι ένα βασικό δικαίωμα η πρόσβαση στη ε, φάρμακα. για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και προσωπικά διαφωνώ κάθετα να υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό. Το θέμα των ατομικών ελευθεριών ήδη νομίζω έχω πει τη γνώμη μου, δεν πρόκειται περί αυτού. Πιστεύω, ελπίζω ότι μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα αλλάξετε γνώμη, αλλά δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτό που έχω ήδη πει. Δεν υπάρχει στο κείμενο και η άκτα δεν αλλάζει το ενοχικό δίκαιο. Αν ένα κράτος μέλος σταματήσει κάποιον στα σύνορά του και ελέγξει, είναι δικαίωμα του κράτους μέλους. Αλλά δεν είναι δικό μου σφάλμα αυτό, ούτε δικό σας, ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην άκτα λοιπόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα ή επιπλέον, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητες. Έπειτα, σε τι χρησιμεύει. Κρίμα που δεν μπορέσατε να είστε παρόν στη συζήτηση αυτή. Γιατί στα τέλη της συζήτησης στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα ανέφερα ένα στοιχείο που σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται είναι η σημασία όλων αυτών για τους εργαζόμενούς μας, τους ερευνητές μας, την οικονομία μας. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι των οποίων η δουλειά εξαρτάται από τα πνευματικά δικαιώματα. Και μιλάμε για την έξοδο από την κρίση και ότι χρειάζονται περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και εδώ λέτε γιατί, σε τι χρησιμεύεται να προστατέψουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτό και ιδιαίτερα όταν προέρχεται από πλευρές όπου λέγονται διάφορα και ποτέ δεν γίνεται αυτή η παρατήρηση για το, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει άκτα στην απασχόληση. επενδύσεις, ποιος μπορεί να υποβάλει τέτοια αίτημα ή καταγγελία. Εδώ θα μείνουμε στα όσα γίνονται για το Trade Defense Instrument. Δηλαδή, οι ε, μπλεκόμενες εταιρείες και έπειτα με την ανακοίνωση θα έρθω ενώπιόν σας τη στιγμή που θα έχει οθετηθεί από το σύνολο των επιτρόπων. Αλλά νομίζω πως δεν θα ήταν σκόπιμο εγώ να εκφραστώ τώρα και να πω πράγματα για μια ανακοίνωση που δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Αμέσως μόλις εγκριθεί είμαι έτοιμος να έρθω στην Επιτροπή σας και να τη συζητήσουμε εις βάθος. Κυρία Ντεσαρνές, εμπιστευτικότητα. Η διαφάνεια που συνδέεται με την εμπιστευτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε ώστε τα κείμενα να δημοσιεύονται. Και το τελευταίο κείμενο, αυτό του Τόκιο, δημοσιεύθηκε τέσσερις μέρες μετά από τις διαπραγματεύσεις. Ολόκληρο το κείμενο. Με εντό εισαγωγικών τι έξι επιφυλάξει που υπήρχαν ή που υπάρχουν ακόμα, τρει από την πλευρά την ευρωπαϊκή και τρει από την αμερικανική. Υπήρξε μια ερώτηση στον Ombudsman για... του ρωτήθηκε αν θεωρεί πως η διαφάνεια θα πρέπει να είναι απόλυτη στις συμφωνίες ή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. και ότι το κοινοβούλιο δεν μπορεί ποτέ να εμπιστεύεται το εκτελεστικό όργανο. Όμως εμπιστεύεστε τον ε, Ombudsman, τον διαμεσολαβητή και είπε ο ίδιος όχι, η Κομισιόν μπορεί να ε, κρατήσει κάποια έγγραφα εμπιστευτικά γιατί διαφορετικά αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική της θέση. Και περί αυτού πρόκειται. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να σας διευκολύνουμε τη ζωή όσον αφορά τις διαπραγματεύσει που κάνουμε. Αλλά τελικά ε, η Κομισιόν είναι που πρέπει να διαπραγματευτεί και δεν μπορώ να θέσω σε τόσο δύσκολη θέση τους διαπραγματεύτέ μου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο αποτελείται από ειδικού στη ΣΑΚΤΑ. Είναι το κύριο θέμα του Κοινοβουλίου, από ό,τι βλέπω. Εμένα μου πήρε μήνες να καταλάβω περί τίνο πρόκειται. Γιατί είναι αρκετά περίπλοκη αυτή η συμφωνία. Έχω την εντύπωση λοιπόν πως για τους ευρωβουλευτές είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι για μας. Μερκοσούρ. Ναι. Ψηφίσατε ένα ψήφισμα. Και αν χρειαστεί να εφαρμοστεί κατά γράμμα αυτό το ψήφισμα, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσει. Ναι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και μάλιστα τα όσα περιλάβατε σε αυτό το ψήφισμα, που είστε ελεύθεροι φυσικά να το ψηφίσετε, δεν ανταποκρίνονται καθόλου στα κριτήρια του ΠΟΕ. Καθόλου μα καθόλου. Τα κριτήρια είναι η υγεία, η υγεία της ανθρωπότητας και έπειτα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες ηθικές παρατηρήσεις, ηθικής φύσης παρατηρήσεις, τις οποίες συμμερίζομαι, αλλά Όλα αυτά δεν εντάσσονται στα κριτήρια του ΠΟΕ, για παράδειγμα για να σταματήσουν κάποιο είδους αγωγές. Και η άποψη που εσείς και ορισμένοι άλλοι έχουν για την αμοιβαιότητα πραγματικά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για οτιδήποτε. Ναι, αλλά κυρία μου, Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να συμφωνούμε με κάτι, να, το, να μας αρέσει και το αν αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, στην πράξη. Όταν πρέπει να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, πρέπει να σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Μα είστε ελεύθεροι να ψηφίζετε ό,τι θέλετε. Να ζητήσετε από την Κομισιόν να σταματήσει κάθε εμπορική διαπραγμάτευση. Μπορείτε να το πράξετε αυτό αλλά οι όροι που θέλετε να μας επιβάλλετε μέσα σε αυτό το ψήφισμα, εντάξει το λαμβάνουμε υπόψη, θα το διαβάσουμε προσεκτικά, θα δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε στην διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το ψήφισμα κατά γράμμα. Το Πακιστάν. Είδατε το μέτρο που προτείνουμε. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση για το Πακιστάν μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ζήτησε να υποβάλουμε πρόταση. Από όσο γνωρίζω, όλα τα κράτη-μέλη αντιπροσωπεύονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ψηλότερο επίπεδο και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Το πακέτο λοιπόν που προτείνουμε είναι ένα πολύ μετριοπαθές πακέτο. Και κανένας δεν συμφωνεί. Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι όχι έπρεπε να προχωράει περισσότερο, αλλά λένε πως δεν πάει αρκετά μακριά. Οι Πακιστανοί διαφωνούν γιατί, διαφωνούν γιατί περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα. Κανένα λοιπόν δεν συμφωνεί και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι τελικά ίσως η πρόταση αυτή δεν να είναι τόσο ανόητη και να ανταποκρίνεται στα όσα είναι δυνατόν να γίνουν μέσα στη σημερινή κατάσταση. Και αυτό είναι που θελήσαμε να κάνουμε. Τώρα αν ο αντίκτυπο θα είναι θετικό, ναι. Θα μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό. Δεν είναι προφανέ το πώ θα το μετρήσουμε όλα αυτά. Γιατί όπως είπε και η κυρία Κουίστο, ότι υπάρχει και ένα πολιτικό στοιχείο μέσα σε όλα αυτά που δεν είναι προφανές να μετρηθεί, αλλά οι αρχική κρατών και κυβερνήσεων είναι αυτοί που αποφάσισαν ότι έπρεπε κάτι να προτείνουμε και το αυτό κάναμε. Αμοιβαιότητα. Ναι, πρόεδρε, το ξέρω, αλλά αφού μου θέσαν τόσε ερωτήσει, τι να κάνω. Προσπαθώ να τι απαντήσω. Αμοιβαιότητα, ναι. Εργαζόμαστε για μια σχετική πρόταση. και έχουμε μια αρκετά ξεκάθαρη ιδέα για το πώ θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά πριν να υποβάλουμε πρόταση, πρέπει καταρχήν να γίνει ε, εκτίμηση αντικτύπου και αυτό παίρνει μήνε. στην πράξη δεν θα μπορέσουμε να σας υποβάλουμε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο πριν το νωρίτερο τον Ιούλιο και πιθανότατα το Σεπτέμβριο του 2011 δεδομένων των προθεσμιών που πρέπει να τηρήσουμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί είναι κάτι αρκετά πολιτικού χαρακτήρα και εγώ θεωρώ ότι είναι κάπως παράξενο να υπάρχει συνένεση και στην Κομισιόν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτή την υπόθεση και έπειτα μόνο και μόνο λόγω προθεσμιών να περιμένουμε νέα μήνες πριν να μπορούμε να σας υποβάλουμε νομοθετική πρόταση είναι ένα μυστήριο. Θα πρέπει μάλλον να ξανασκεφτούμε αυτή τη διαδικασία που είναι όμως ε, καθιερωμένη και μάλιστα σε κάθε συζήτηση μου ζητάτε άλλη μια εκτίμηση ε, αντικτύπου. Κύριε Ζαντό. Για την Εθανόλη. Σίγουρα δεν είναι μεγάλη χώρα παραγωγός του Πακιστάν. Θα σας πω όμως το Όλοι μας ασκούν κριτική γιατί μιλάνε για το γεγονός πως έχουμε μόνο υφαντουργικά. Ναι, όμως οι εξαγωγέ από το Πακιστάν είναι κυρίως υφαντουργικά. Έχουμε λοιπόν τοποθετήσει και κάποια προϊόντα που δεν είναι υφαντουργικά σε αυτόν τον κατάλογο για να μην νομίζει κανείς πως στοχεύουμε μόνο σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Και να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάναμε και γιατί. Μιλάμε για περιορισμένες καταρχήν ποσότητες. Σας είπα πως μόλις ετοιμαστεί η ανακοίνωση θα έρθουν σας την παρουσιάσω. Οι εξαγωγικές δομές ποτέ δεν κατάλαβα, για παράδειγμα, γιατί πρέπει να κατηγορήσουμε τη Γερμανία που κάνει τόσες εξαγωγές. Εγώ το θεωρώ τα παράξενο να ασκούμε κριτική ε, στο κράτος μέλος που είναι ο πρωταθλητής των εξαγωγών. Μα δεν νομίζω πως χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και για τα όσα είπατε για τις κλιματολογικές αλλαγές, εμείς το προσέχουμε το κλίμα και είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε υπόψη. Και για τον κύριο Σόλτς, για τα ΤΕΚ, έχουμε πρόγραμμα έτσι ώστε να κάνουμε κάποιους προβληματισμούς από κοινού για τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις, για τη χρηματοδοτική κρίση, για την ανάκαμψη και ανάταξη της οικονομίας, για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση και όλα αυτά θα δούμε την ε, καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, την δημιουργία της βάσης αυτής της διατλαντικής αγοράς και θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες ελπίζουμε έτσι ώστε να έχουμε κάποια παραδοτέα και σε αυτό τον κλάδο ε, σύντομα να σας παρουσιάσουμε. Για τα όσα μας είπε ο κύριος Ντάρτμουτ, Σας εξήγησα και πριν ποια είναι η άποψή μου για το θέμα αυτό και για τα τρία έτη. Νομίζω ότι τα καταλάβατε για τις γεωργικές επιδοτήσεις και αν υπάρχει θέμα dumping εδώ, νομίζω ότι στο παρελθόν ναι, σίγουρα. Αλλά πιστεύω πως οι περισσότερες επιδοτήσεις τώρα προέρχονται από το Green Box που δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει τρευλώσεις. Δεν λέω πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι από τους μεγάλους εξαγωγείς γεωρικών προϊόντων σίγουρα εμείς δεν είμαστε χειρότεροι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις προσπάθειες που κάνετε να απαντήσετε στις τόσες ερωτήσεις που ακούσατε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μείνετε λίγο λεπτά ακόμα, γιατί πραγματικά λυπάμαι που τρεις συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Θα τους δώσω το, λόγο για ένα λεπτό και μετά θα σας δώσω και δύο λεπτά να τους απαντήσετε. για να μην ε, αργήσουμε υπερβολικά πολύ. Ο κύριος Ντεζίρ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις σύντομες ερωτήσεις, κύριε Επίτροπε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν έχουμε καλύτερες εμπορικές σχέσεις και πιο ισορροπημένες μεταξύ Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ε, Πού θα καταλήξουμε, τι γίνεται με τη μάχη του Ουάν. Και για τα νομισματικά θέματα, μήπως θα έπρεπε να το δείτε και εσείς και ο Ερμόδιος Επίτροπος και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν υπάρχουν κάποια εμπορικά, θέματα, ε, εμπορικά επιχειρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποκαταστήσουμε τις ισοτιμίες για την αμοιβαιότητα. Εδώ μπλέκουμε δύο συζητήσεις. Καταρχήν το ότι δεχτήκαμε μη συμμετρικό άνοιγμα αγορών από τις αναπτυσσόμενες αγορές, δηλαδή το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και επίσης θα δούσε συνέχεια στο γύρο της Ντόχα, που ζητάμε λιγότερα από ό,τι μας ζητάνε. Και έχουμε βέβαια και το θέμα των ε, κρατικών των δημοσίων προμηθειών. Ωραία. Για την αγορά λοιπόν αυτών ε, νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε και κάποια περιθώρια στις εθνικές ρυθμίσεις, στις εθνικές κυβερνήσεις, γιατί υπάρχει και το θέμα των υπηρεσιών κοινή ωφελία. Αμοιβαιότητα, πολύ σωστά. Τι σημαίνει αυτό όμως, θα απαρνηθούμε η παράδειγμα η τιμολόγηση του ύδατος ή της ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται από το κράτος. Μας είπατε ότι θα παρουσιάσετε και μία ανακοίνωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τα, την κλιματολογική αλλαγή. Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων θα το τοποθετήσετε, γιατί έχουμε την ανακοίνωση για το εμπόριο και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε και τα θέματα αυτά. Ο κύριος Ρινάλντι έχει το λόγο. Thank you, I... Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα την συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για το Πακιστάν και δεν έχω καταλάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταρχήν, αφήνω την άκρη, στην άκρη στο παλιά και λέω ότι στηρίζουμε. Εντάξει, το στηρίζουμε. Λοιπόν, αλλά δεν έχω καταλάβει, επανέρχομαι, στο κατά πόσο... έχουμε εδώ ένα πακέτο μέτρο ένα πακέτο μέτρων το οποίο με κάποιο τρόπο να αντισταθμίζει τις τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το ίδιο το πακέτο στον ε, κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας. Έχετε σκεφτεί πώς το πακέτο αυτό μπορείτε να εντάξετε κάτι που να τους βοηθήσει. Για το άκτα εντάξει, το μόνο που έχω να πω είναι πως υπάρχει προφανής ε, ανησυχία πως οι γεωγραφικές ενδείξεις θα είναι πολύ λιγότερο προστατευτικές από τα εμπορικά σήματα τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές και αυτό θα σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και αυτό μας ανησυχεί Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να το θίξουμε. Και τέλος, ο κύριος Ένστρομ, πράσινη. Μία ερώτηση για τις γεωγραφικές ενδείξεις και το άκτα. Μιλήσατε για πλήρη απόρριψη ε, ε, των θέσεων αυτών από τις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό φαίνεται και από την ίδια τη συμφωνία. Κοιτάξτε, παράγραφο 1.3.2 που λέει αυτή η συμφωνία, αυτή η συμφωνία αυτή δεν, απορρέ, δεν, αυτή η συμφωνία αυτή δεν, απορρέα, δεν απορρέει ούτε μία υποχρέωση να επιβληθούν κυρώσεις κτλ. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν πως οι γεωγραφικέ ενδείξει δεν προστατεύονται στι ΗΠΑ. Άρα λοιπόν εντάξει. Εκτός λοιπόν έμειναν, αλλά μας είπατε πως έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, φαίνεται οι γεωγραφικές ενδείξεις τελικά να είναι εντός της συμφωνίας. Μπορείτε να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Ευχαριστώ. Που έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε σε αυτές τις τελευταίες ερωτήσεις. Να ξεκινήσω λοιπόν με την τελευταία ερώτηση για την άκτα. Δεν είναι η συμφωνία η οποία αλλάζει το ενοχικό δίκαιο, άρα λοιπόν για τις γεωγραφικές ενδείξεις δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. για οποιαδήποτε από τα συμβολόμενα μέρη. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε εδώ την νομοθεσία περί γεωγραφικών ενδείξεων στη ΣΥΠΑ. Όμως, στοχεύει η συμφωνία αυτή στην επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Και εδώ προσφέρουμε την ίση μεταχείριση σε όλους τους κατόχους αυτών των δικαιωμάτων, όπως επίσης και για τις γεωγραφικές ενδείξεις, κάτι το οποίο απέρριψαν στην αρχή, αλλά μετά δέχτηκαν. Άρα λοιπόν μπορούμε να το επιβάλλουμε μέσω αυτού. Μόνο στις χώρες όμως όπου αναγνωρίζονται οι γεωγραφικές ενδείξεις. Αυτό έχουμε τοποθετήσει στην συμφωνία. Είναι η επιβολή λοιπόν αυτού του του δικαίου. Και όταν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία, βεβαίως είναι αδύνατο να επιβληθεί. Στην πράξη λοιπόν, η ενησυχίε για τη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, όπου έχουμε το Εθνικό Μητρό, προστατεύονται οι γεωγραφικές ενδείξεις και όπου θα μπορούσε να γίνει επιβολή στα σύνορα, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνετε τη διάκριση μεταξύ του τελικού χρήστη και τα προϊόντα σε καθεστώς διαμετακόμισης. Εσείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιτύχετε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιτύχουμε την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων και αυτό πρέπει να το κάνετε και εσείς ως κράτη-μέλη, αλλά πολλά κράτη δεν το δέχονται. Το εξήγησα αρκετά σαφώς, ελπίζω. Για τον κύριο Ρινάλδη, αντιστάθμιση Άκουσα τι είπατε στην ε, Ολομέλεια. Θα δούμε αν είναι λοιπόν ε, δυνατό αυτό ή έχει και για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Σας έδωσα μία απάντηση. Αναγνώριση μερική γιατί αρκετά κράτη, επαναλαμβάνω, δεν θέλουν την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό που δεν αληθεύει είναι ότι ω αποτέλεσμα τη άκτα θα χάσουμε ε, θέσεις Μα δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυξάνουμε το ε, ποσοστό προστασία. οπότε σε αυτό που είπατε το ήταν αντιφατικό. Η μάχη των ισοτιμιών, αν θα πάρουμε εμπορικά μέτρα, όχι αυτή τη στιγμή. Με ρώτησαν και στην Ολομέλεια αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάποια πρόταση για να λάβουμε εμπορικά μέτρα όπως ε, σκέφτονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί εκεί το Κογκρέσο ψήφισε ένα κείμενο, το οποίο βέβαια πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία. Είναι και το θέμα το προς ποια κατεύθυνση θα κλείνει ο πρόεδρος των Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει πρόκειται για ένα απλό ψήφισμα στι ΗΠΑ, δεν είναι νόμος. Εμείς παρόμοια σκέψη ακόμα δεν κάνουμε. Και για τις δημόσιες προμήθειες, εδώ έχουμε και τις υπηρεσίες κοινή ωφελία. Αυτό είναι πρόβλημα, α, όχι μόνο εμπορικό. Έχουμε και τη σχετική οδηγία, αρκετέ μάλιστα οδηγίε. Έχουμε την οδηγία που είναι υποσυζήτηση. Να δούμε λοιπόν ποιε θα είναι οι εμπορικέ συνέπειε. Τώρα για την κοινωνική και τις κοινωνικές επιπτώσεις προσπαθήσαμε να εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην ανακοίνωση. Νομίζω όταν μιλάτε για κοινωνική ευθύνη έχετε στο νου και την ανάπτυξη. Έχω λοιπόν στόχο να εκδώσουμε μία ανακοίνωση συγκεκριμένα για το εμπόριο και το ρόλο που έχει στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων ε, κρατών, ε, χωρών, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά. Ενδιαφέρουσα και πλούσια συζήτηση. Ίσως την επόμενη φορά θα πρέπει να περιορίσουμε κάπως τα θέματα. Να σας διαβεβαιώσω πως δεν σας ζηλεύουμε που είστε στη θέση αυτή. Ούτε θα θέλαμε να πάρουμε τη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ να σας κάνουμε ερωτήσεις. Για να ξέρουμε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Και για τις προσπάθειες που κάνετε και τις απαντήσεις που μας δώσατε.